Mes chers collègues, je vous demande de prendre place. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε για να δούμε το σημείο 21α. Να δώσω το λόγο στον Τόμας Μαν για να δούμε πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις για τις υπηρεσίες στα αεροδρόμια. Σας προειδοποιώ, η συνεδρία θα είναι δύσκολη και είναι ένα σημείο που θα απασχολήσει και την Επιτροπή Μεταφορών. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να βελτιωθεί και η φωνή σας. Να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση για τα ζητήματα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει από κοινού με την Επιτροπή Μεταφορών σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση εδάφους υπήρξε μια συνάντηση των σκιωδών εισηγητών της Επιτροπής Μεταφορών όπου ήμουν παρόν και εγώ παρουσίασα τη θέση της δικής μας Επιτροπής. Ο και κ. Τσαζάνα έκανε μια νέα πρόταση που περιλαμβάνει και ορισμένε συμβαστικέ λύσει που έχουν τύχει συζήτηση προηγουμένω. Πρόκειται για το εξή: Ότι πρόκειται να πρέπει να υπάρχει ένα τρίτο πάροχο για ορισμένα αεροδρόμια, μεγάλα αεροδρόμια, αλλά έχει αυξηθεί το κατόφλι. 15 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ η Κομισιόν είχε προτείνει μόνο 5. Και αν το, τα εμπορεύματα ξεπερνούν τις 200.000 τόνους και όχι μονάχα 100.000 τόνους, τότε σε αυτή την περίπτωση απαιτείται να υπάρχει ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών, μια μεγαλύτερη φιλελευθερωποίηση. Η εναλλακτική <clears throat> λύση είναι να υπάρξει μια λύση, μια λύση επικουρικότητα ουσιαστικά, δηλαδή το κάτω μέλο να είναι αρμόδιο να αποφασίσει αν πρέπει να υπάρχει ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών ή όχι. Όσω μπορεί να υπάρξει λοιπόν μια συμβαστική λύση από τη βάση αυτή. Ένα τρίτο θέμα είναι πότε θα τεθούν σε εφαρμογή όλα αυτά. Η πρόταση ήταν πέντε χρόνια μεταβατική περίοδο συν δύο προς 7 χρόνια, δηλαδή ε, ε, 7 χρόνια μεταβατικό διάστημα. Περισσότερη φιλελευθερωποίηση από τη μία πλευρά σημαίνει ότι θα πρέπει να διατηρηθούν και αυτά τα οποία έχουμε αποφασίσει εμείς ως Επιτροπή ε, κοινωνικών θε, θε, θεμάτων. Επομένως, αυτό το οποίο έχουμε εμεί ζητήσει σε επίπεδο συμβαστικού, επιπέ, ε, επίπεδου να παραμείνουν οι κοινωνικές διατάξεις, να υπάρχει ένα μακρύτερο χρονικό διάστημα κατάρτισης των εργαζόμενων σε υπηρεσίες ε, εδάφου, επίσης να παραμείνουν τα, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή ως πάροχοι και επίσης να αντιμετωπιστεί το θέμα της κατάρτισης όπως είπα. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι ανοιχτό είναι ότι ορισμένοι ισχυώδεις εισηγητές, όχι όλοι, είπαν ότι θα πρέπει ίσως να αλλάξουμε την παράγραφο 12, πρόκειται για το εξή. Οι κανονισμοί που εμείς έχουμε ε, δημιουργήσει αφορούν τις ε, βαλίτσες, το, τα εμπορεύματα την ε, εξυπηρέτηση με καύσιμα και τις άλλες συναφείς υπηρεσίες για τα αεροπλάνα. Μόνο αυτά είναι στοιχεία που μας ενδιαφέρουν. Σε όλα τα άλλα στοιχεία υπάρχει απόλυτη φιλελευθεροποίηση και λειτουργεί εδώ και πολύ καιρό ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πρόβλημα γιατί μήπως θέλουμε να διευρύνουμε τον τομέα ε, εφαρμογής αυτού του κανονισμού να έχουμε όλους τους τομείς, τους 11 τομείς οι οποίοι θα καλύπτονται από την τελική λύση. Δεν ξέρω λοιπόν αν αυτό θα μπορέσει να μας οδηγήσει σε μια κοινή λύση. Εγώ προσπαθώ να διερευνήσω κατά πόσο αυτό είναι δυνατό. Την επόμενη εβδομάδα κάποιες πολιτικές ομάδες θα λείπουν από τις Βρυξέλλες, επομένως δεν μπορούμε να έχουμε σκιώδεις συζητητές από αυτούς. Θα έχουμε μονάχα κάποιες διμερείς επαφέ. αλλά στο Στρασβούργο εγώ θέλω να κάνω μια συνάντηση με όλου του σκιώδεις συζητητές για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κοινή γραμμή. Επίσης, <clears throat> η χρονική ε, αλληλουχία είναι σημαντική. Μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου θα πρέπει, αν θέλουμε στα μέσα Φεβρουαρίου να έχουμε μια κοινή λύση, θα πρέπει να επενδύσουμε και περισσότερο χρόνο για να υπάρξει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, όποιος δεν θέλει κανένα κανόνα, όπως είπαν ορισμένες πολιτικές ομάδες, δεν πρόκειται να αποφασίσει τίποτα. Αλλά υπάρχουν τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τα, εμπορεύματα, τα, τις χρονοθυρίδες και την προστασία από, από την ε, ηχορύπανση. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά λοιπόν, εν συντομία, ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να καταλήξουμε σε μια τέτοια συμβιβαστική λύση η οποία να μπορέσει να γίνει δεκτή από όλους και να δημιουργήσουμε ένα κοινό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλο αυτό λόγο. Εγώ θέλω απλώς να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων ότι, όπως είπε ο κύριος Μαν, είναι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή Μεταφορών και θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή τη δυνατότητα να καταθέσουμε και πάλι τις τροπολογίες μας στην Ολομπέλεια αν η συμφωνία η οποία θα εξευρεθεί δεν θα φαίνεται ικανοποιητική. Σας ευχαριστώ λοιπόν κυρία Μαν. Μήπως θέλει να λάβει το λόγο η Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Υπάρχει κάποιος από την Κομισιόν. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ κυρία μου. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα λάβω το λόγο εν συντομία γιατί ξέρω ότι είναι πεφορτωμένη η ημερήσια διαταξή σα. Θέλω να τονίσω το γεγονός ότι η Κομισιόν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να υπάρξει αυτό το κείμενο για την εξυπηρέτηση σε ενδιάμεσους σταθμούς, γιατί χωρίς αυτή τη ρύθμιση το κείμενο του 2006 θα μείνει ως έχει. Εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια βελτίωση στα θέματα αυτά. Η Κομισιόν έχει σαν στόχο να βελτιώσει την κατάρτιση του προσωπικού που ασκούν αυτή την εξυπηρέτηση και το δικό σας μήνυμα είναι ιδιαίτερα σαφές για το ότι εμεί θα πρέπει να επιμείνουμε πολύ περισσότερο για τα σημεία αυτά, κάτι το οποίο το δέχεται η Κομισιόν. Επίση, για να εξασφαλίσουμε καλύτερη λειτουργία των αεροδρομίων με ελάχιστα πρότυπα ποιότητο, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο σήμερα να το επιτύχουμε. γιατί αυτό θα έχει και επιπτώσεις στις συνθήκες με τις οποίες μεταφέρονται οι επιβάτες και επίσης θα οδηγήσει και σε προβλήματα σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών εξυπηρέτησης που θα πρέπει να παρέχουν την καλύτερη υπηρεσία για το χαμηλότερο τίμημα προς τους επιβάτες. Το Κοινοβούλιο έκανε ιδιαίτερα σαφές το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει φιλελευθερωποίηση και άνοιγμα της αγοράς. Για τα θέματα αυτά, ακόμα και αν εμείς Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει ένα τρίτο πάροχο υπηρεσιών εδάφου για τα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε το θέμα των κατοφλίων και επίσης το θέμα των μεταβατικών χρονικών περίοδων. Και για το θέμα αυτό η Κομισιόν είναι έτοιμη να ακολουθήσει την γραμμή του Κοινοβουλίου διότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ πολύπλοκο για το θέμα εξάλλου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό των δικαιωμάτων και, των, και της μεταφοράς των δικαιωμάτων από μία εταιρεία σε μία άλλη. Εκεί που αναφέρονται λοιπόν τα θέματα αυτά και επίσης το άρθρο 40 που είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τη δικαιοδοσία των κρατών μελών για τα θέματα αυτά και εμείς θέλουμε να ακούσουμε την άποψη του Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στο κείμενο αυτό ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την υπηρεσία, τις υπηρεσίες που παρέχονται στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συνεκτική δέσμη μέτρων για την ηχορύπανση, για τις χρονοθυρίδες και για την εξυπηρέτηση εδάφους, ώστε να ενισχύσουμε τη θέση των ευρωπαϊκών αεροδρομίων στον διεθνή ανταγωνισμό. Σας ευχαριστώ. Όπως καταλαβαίνετε η Επιτροπή μας δίνει μεγάλη σημασία στο να υπάρξει η σωστή αντιμετώπιση του προσωπικού εδάφους και της, ε, του σεβασμού των ε, συμβολέων τους. Αλλά φυσικά πρέπει να ληφθεί υπόψη και το θέμα του ανταγωνισμού. Θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες τώρα. Εάν συμφωνείτε, έχει, υπάρχει πλήρης παρουσία από τις πολιτικές ομάδες. Περιμένουμε ένα-δύο λεφτά. Από τα Συνάδελφοι, αν θέλετε να ξεκινήσουμε. Σημείο 22. Στο σημείο 22, η έκθεση της κυρίας Λόπε Φοντανιέ, παράγραφος 1, νέα, 48, υπέρ. Κατά. Αποχές για να επαληθεύσουμε. Εψήφισαν άπαντες πέρασε τη ψηφοφορία. 17 υπέρ 17 κατά λέει πρόεδρος δεν εγκρίνεται 50 τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Επαληθεύουμε για την 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες πέρας. 16 προς 18. Δύο δεν εγκρίνεται. Κύριε Ρή, Δεν λειτουργεί η κάρτα μου νομίζω. Στη... Από τη σωστή πλευρά. 51. Καταπίπτει. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55. Μπαχ. Υπέρ.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 κατά, αποχές, απορρίπτεται. 61 υπέρ, συγγνώμη, 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική G, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική KK, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική, συγγνώμη, τροπολογία 71 υπέρ. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική JJ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 83 και 172 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική I υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 101 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Χωρίς τους όρους και μηχανισμοί του. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 4 υπέρ. Ρέτζι 4 υπέρ. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική N. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική M. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική O υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η φιλελεύθερη είναι υπέρ. 122 υπέρ. Ε, εντάξει, να επαληθεύσουμε για το 122. Επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. είναι οι σοσιαλιστές υπεράριθμοι. Υπάρχει ένας παραπάνω. Είναι υπεράριθμοι κατά έναν βουλευτή. Σέργιο, σας παρακαλώ, βγάλτε την κάρτα σας. Πέρας. Εγκρίνεται. 25 προς 17 με μία αποχή. Είχα δίκιο. 122 υπέρ. Κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτζι 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 123. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική π. Όχι, όταν η φιλελεύθερη είναι υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική π. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 129 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. 130. Υπέρ. Κατά αποχέ, απορρίπτεται. 131. Υπέρ. Κατά απόχέ, απορρίπτεται. 132. Υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 135. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 134. Υπέρ. Με συγχωρείτε. 133. 133. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέτζι 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική Q υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 143 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Ρέτζι 11 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική R υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική S υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 148 υπέρ κατά απόχέ, απορρίπτεται. 149 υπέρ κατά Αποχέ. απορρίπτεται. 150 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 151. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτζε 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτζι 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτζι 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτζι 6. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. Ρέτζι 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 154. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 155. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. 156. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 157. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική ΤΑΒ Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 160. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 162. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική γιού, Υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνεται 166 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 167, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 168 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 169 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. «170 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική W υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 175 υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να σηκώνετε τα χέρια παρακαλώ. 180 υπέρ. Κατά. 180 πουρ. Ε, συγγνώμη. Υπέρ. Κατά αποχές να επαληθεύσουμε. Εψήφισαν άπαντες. Εντάξει, πάνε όλα καλά. Πέρα τη ψηφοφορία. 39 υπέρ, 7 κατά. Πραγματικά ήταν απαραίτητο να επαληθεύσουμε, εγκρίθηκε. Δεν ήταν σαφές. Με προφορική τροπολογία, για να τέσσερα στο χειρός. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 185 υπέρ. Κατά. Α, υπέρ 185. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία του εισηγητού. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 191 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται. Συμβαστική A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για τι φυτογλυκές αναφορέ. 2 υπέρ κατά Υπέρ του 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Με προφορική τροπολογία. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επαλήθευση. Επαλήθευση για το 3. Και πάλι είναι υπεράριθμοι στους σοσιαλιστές. Περισσεύει ένας. Πέρα στις προφορίες. 18 υπέρ, 27 κατά. Δεν εγκρίνεται, είχατε δίκιο. 4 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 με προφορική τροπολογία. Καταπίπτει 8 υπέρ Κατά αποχές απορρίπτεται. Μην πανικοβάλλεστε. 9. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 12 est tombé parce qu'il était couvert, donc je pense que le 12... Νομίζω ότι και η 12 καταπίπτει. Η προηγούμενη πάντως καλύπτωταν από την προηγούμενη. Συμβαστική D, υπέρ. Κατά, απόχέ εγκρίνεται. 15, υπέρ. Κατά, απόχέ εγκρίνεται. 16, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεκαεπτά υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Με συγχωρείτε. 17 δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε γιατί 166 δεν ψηφίζουμε την 17 γιατί η 166 εγκρίθηκε. Θα ψηφίσουμε όμως την 18 διότι απορρίφθηκε 168. 18 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. Συμβαστική B. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. αποχέ Εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. αποχέ Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. αποθέσει, Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Συμβαστική ΣΥ. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 36. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Υπέρ τη 36. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. F υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Ετυλογική σκέψη 14 στα Κατά Καταπίπτει ε. Υπέρ. Υπέρ τη συμβιβαστική ε. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 45. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. 197 υπέρ. Κατά απόχε εγκρίνεται. 100 απορρίπτεται, συγγνώμη. 198 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 199 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική Z υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AA υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 205 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 207 Να μην την ψηφίσουμε. Σας προτείνω να μην την ψηφίσουμε. Συμφωνούν οι ομάδες. 210 υπέρ. κατά, αποχές, απορρίπτεται. 208 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 211 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική BB υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 213 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 214 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 215 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 216 υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβαστική CC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική DD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 220 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 223 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε την 223? Ας επαληθεύσουμε την 223. Ε, 18 προς 24 κατά τρεις αποχές. Είχε δίκιο κυρία Μωρά. Δεν εγκρίνεται. 223 υπέρ. Με συγχωρείτε, 224 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 225 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 226 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 227 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 228 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 229 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ή ε, ε, ΕΕ. υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. FF υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. GG υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 235 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 236 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 238 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 237 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 239 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 240 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 241 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 242 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 243 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 244 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 245 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. Συμβιβαστική HH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 248 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική II υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 251 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 253 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 254 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 255 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 256 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το κείμενο στην τελική φάση. Είναι υπεράριθμο το ΕΛΚ. Εψήφισαν άπαντες πέρας. 39 υπέρ, 5 κατά. Συγχαίρουμε, συγχαίρουμε την εισηγητρία μας. Et Σας ευχαριστώ κυρία Λόπε Φοντανιέ. Μάλλον να της μεταβιβάσετε το μήνυμα, διότι δεν μπορούσε να είναι μαζί μας σήμερα το πρωί. Δέχτηκε όμως για την εύρυθμη Εξαγωγή της ψηφοφορία να ψηφίσουμε απόψε, σήμερα το πρωί. Συνάδελφοι, στην Επιτροπή Δημοσιονομικών και Οικονομικών Υποθέσεων το θέμα αυτό τελικά δεν συζητήθηκε, οπότε το δικό μας κείμενο θα περάσει στην Ολομέλεια. Απορρίφθηκε η έκθεση Φερέρα στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση μέχρι να περάσει η έκθεση της κυρίας Λόπε Φοντάνιε στην Ολομέλεια. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα τώρα. Ευχαριστώ λοιπόν την εισηγητριά μας που μας ε, επέτρεψε να φτάσουμε σε αυτήν την τοποθέτηση. Ερχόμαστε τώρα στο σημείο 23 για την ευθύνη του κράτους σημαίας σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ των, των εταίρων. Άρθρο 1. Σας προτείνω να ψηφίσουμε από κοινού τις τροπολογίες 1, 2, 4. Συμφωνείτε ψήφι υπέρ κατά αποχές. Δεκτές τροπολογία 4 και τρανς 5 υπέρ κατά αποχέ αδεκτέ 5 και τρανς 6 όχι όχι είναι χωριστές 5 κατά Χε. δεκτή τρανς 6 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Πέρας ψηφοφορίας. 21 υπέρ 3 κατά. 21 υπέρ 23 κατά, συγγνώμη, απορρίπτεται. 6 και 7 μαζί, αν δεν έχετε αντίρρηση, ψήφι υπέρ. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, σε. Ναι, λέξουμε. Δεν βλέπω. Δεν εκρίθη. Εκπίπτει η 8. Τραν 7 ψήφι υπέρ. κατά αποχές δεχτεί Οκτώ και τραν εννέα. υπέρ κατά αποχές δεχτεί τροπολογία εννέα. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά ας δούμε, ας ελέγξουμε για την εννέα. ψήφισατε Ψήφισατε όλοι, πέρας. 21-23 απορρίπτεται. Μεταφορές 10 υπέρ. Κατά ποχές δεκτές. Δεκτή. 10 και μεταφορές 11 υπέρ. Κατά ποχές δεκτές. 11 υπέρ. Κατά θα ελέγξουμε για την 11. Άρχεται. Πέρασε. 26 με 18 εγκρίνεται. 12 μεταφορών, 12 μάλλον και 13 μεταφορών υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνονται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Μεταφορές 15 υπέρ. Κατά. Ψηφίστε καλύτερα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 15 υπέρ. Κατά Απόχε. Να ελέγξουμε για τη 15. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Πέρας. 21-23. Απορρίπτεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, θα σε ελέγξουμε. Πέρας. 26-17 εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 17 εγκρινεται Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 και 14 μεταφορές υπέρ. Αποχές δεκτές. 21 και 16 τρανσπορ υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. 22, 72 και 17 μεταφορών υπέρ κατά δεκτές. 23 της εισηγητρίας και 18 μεταφορών υπέρ κατά αποχές δεκτές. 24 και 19 μεταφορών υπέρ κατά αποχές δεκτές. 25 και 20 μεταφορών transport 34 pour. 34 μεταφορών υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 34. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 20-23 απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά αποχέ ε, κρίνεται. 26 και 21 μεταφορών υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 27 και 22 μεταφορών υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 28 και 23 μεταφορών υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνονται. 29 και 24 μεταφορών υπέρ, κατά αποχές δεκτές, 30 και 25 μεταφορών υπέρ, κατά αποχές δεκτές. Μήπως μπορούμε να ψηφίσουμε όλη τη σελίδα Συμπούρμπουλη μέχρι την 31 μεταφορών. Από κοινού όλες μαζί ψήφ υπέρ κατά αποχές δεκτές όλες αυτές τις τροπολογίες. Από την 37 μέχρι την 41 μεταφορών όλες μαζί υπέρ κατά άποχες δεκτές. 46 ως 61 όλες μαζί υπέρ. Όχι, δεν θέλετε. Amendement 46 qui est pour. 46 υπέρ. 46 υπέρ. ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 20 29 21 47. Τα ίδια, ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 21-23. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Πάλι ηλεκτρονικά θα κάνουμε. Υπέρ. Μάλλον έρθει η ψηφοφορία. Πέρασε. 21 με 22. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 49. Όχι, δεν την ψηφίζουμε. Ναι, δεν την ψηφίζουμε. 50. Υπέρ. Θα ελέγξουμε. 50 ηλεκτρικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 22-21 εγκρίνεται. Εγκρίνεται, εγκρίνεται είπα. Εγκρίνεται, δεν είπα δεν εγκρίνεται. 51 είπε. Κατά αποχές θα ελέγξουμε πάλι. 51 ηλεκτρονικά. Πέρασε. 2022 22 λόγω ισοψηφίας απορρίπτεται. 52. Ηλεκτρονικά. Άρχεται. Φωτίσατε, <coughs> ψηφίσατε όλοι πέρας. 22-22 το ίδιο αποτέλεσμα. 53. Ηλεκτρονικά. Ευτυχώς είχαμε πολλή συζήτηση πριν φτάσουμε στην πληροφορία. Πέρασε. 22-22 απορρίπτεται. 54. Άρχεται. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά αποχές θα ελέγξουμε την 55 ηλεκτρονικά. είναι 21-23 απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Για 57 άρχεται. Πέρας. 21-23 απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές θα έλεξουμε την 59. λιγο τικλο τύκλο. Πέρας. 25-19 γίνεται δεκτή. 59 ψηφίζουμε. Όχι, το ξανακάνουμε τότε. Δεν ψηφίσαμε την 58 γιατί δεν είναι κρίση 55, οπότε ψηφίσουμε την 59 και κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Η συγκίτρια την υποστηρίζει, όπως ξέρετε. Πέρασε. 35 με 8 γίνεται δεκτή. 60 υπέρ κατά αποχέ προς το απορρίπτεται αλλά θα επαληθεύσουμε 60 πέρασε 21-22 απορρίπτεται 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Απόχες θα ελέγξουμε για την 63. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 21-23 απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές δεκτή μεταφορές 42 υπέρ κατά αποχές <coughs> εγκρίνεται μεταφορές 1 υπέρ κατά υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε μεταφορές 1 vote 23 με 20 εγκρίνεται. Μεταφορές 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μεταφορές 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το σχέδιο έκθεσης όσο έχει τροποποιηθεί ηλεκτρονικά. Αρχιτεί ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 37-2 εγκρίνεται με 5 αποχές. Το νομοθετικό ψήφισμα άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας 37-2 με 5 αποχές πάλι, το ίδιο αποτέλεσμα. Εγκρίνεται. Και μετά από την απόφαση των συντονιστών θα εφαρμόσουμε τον νέο κανόνα 70, το άρθρο 70 του κανονισμού που μας υποχρεώνει για να δούμε αν συμφωνείτε για, αν για να ανοίξουμε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Αυτό είναι και η έγκρισή σας για να δημιουργηθεί η ομάδα διαπραγματεύσεων από την εισηγήτρια, από τον κύριο Ορή από το ΕΛΚ, τον κύριο Ντεμπάκ από τους Φιλελεύθερους, του, από τον κύριο Λάμπερ για τους πρασίνους. Η κυρία Λάμπερ για τους πρασίνους, συγγνώμη, συγγνώμη. Και, και του κυρίου Λεϊαρίκ για την Γκουε. Οπότε, εγώ θα είμαι και πρόεδρος αντιπροσωπείας και εισηγήτρια. Αν δεν έχετε αντίρρηση, αν έχει τώρα μια ομάδα αντίρρηση, δεν έχω κανένα πρόβλημα να αναλάβει κάποιο την προεδρία της ε, αντιπροσωπείας. Συμφωνείτε? Λοιπόν, ψηφίζουμε για την σύνθεση της αντιπροσωπείας ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη, ο κύριος Λεγιαρίκα έχει το λόγο. Θα σας δώσω το λόγο και μετά την ψηφοφορία, με θέλετε. Μετά θα μου δώσετε το λόγο. Μέσα στην ψηφοφορία δεν μπορώ να σας δίνω το λόγο. Μα τώρα είναι πριν από την ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Λεγιάρικ. Εντάξει, ακυρώνουμε ψηφοφορία. το λόγο. Εγώ συμφωνώ με την έκθεσή σας και την υποστηρίζω, αλλά θεωρώ από την άλλη πλευρά ότι πρέπει να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν για τα θέματα αυτά. Για λόγους αρχής θεωρώ ότι η εφαρμογή του άρθρου 70 σημαίνει ότι η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα έχει το δικαίωμα συζήτησης. Θα κάνουμε λοιπόν μια συμφωνία η οποία λαμβάνει χώρα πριν από τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Για τους λόγους αυτούς εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω την εφαρμογή του άρθρου 70. Αλλά έτσι θα καταψηφίσετε επειδή είναι και η πρώτη φορά που εφαρμόζουμε το άρθρο 70 στην Επιτροπή μας, θέλω να σας απαντήσω με δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατηρήση λέει ότι στην πραγματικότητα σήμερα ουσιαστικά επικυρώνουμε μια τρέχουσα πρακτική της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, δηλαδή επί τη βάση της έκθεσης η οποία είχε εγκριθεί στην Επιτροπή μας, να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις ώστε να επιτευχθεί συμφωνία ή δυνατόν πρώτης ανάγνωσης με το Συμβούλιο. Αυτό καλύπτει και το τροποποιημένο άρθρο 70 του κανονισμού μας. Αυτό το οποίο αλλάζει τώρα στο άρθρο 70 είναι ότι εάν εάν δεν συμφωνούμε να ανοίξουμε διαπραγματεύσει, γιατί φυσικά μπορούμε πάντα να στήσουμε να πάμε πρώτα στην Ολομέλεια και μετά να ανοίξουμε την ε, διαπραγματεύση, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε. Τα ξαναλέω πάλι γιατί τα μπέρδεψα. Το 70 τροποποιημένο. Ουσιαστικά εφαρμόζει την πρακτική της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής που συνίσταται στο εξή. Ότι δεν πρέπει να γίνει τελική ψηφοφορία για το θέμα αυτό, το οποίο ήταν αντικείμενο μιας έκθεσης και αυτό θα πρέπει να πάει στην Ολομέλεια. Αυτό γινόταν για το πακέτο εποπτικών μέτρων. Αυτή ήταν η διαδικασία τη Επιτροπή Νομισματικών και Οικονομικών Θεμάτων να ψηφιστούν όλε τι τροπολογίε και μόνο μετά στην Ολομέλεια να ψηφιστεί το σύνολο τη εκθέσεω και το νομοθετικό κείμενο για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει. Εμεί ποτέ δεν το κάνουμε αυτό. Ίσως στο μέλλον θα πρέπει να το κάνουμε αν θεωρούμε ότι από πολιτική έποψη είναι απαραίτητο να γίνεται κάτι τέτοιο αλλά στην τρέχουσα περίπτωση αυτό το οποίο κάνουμε είναι να έχουμε μια επίσημη επισημοποίηση με ψηφοφορία της πρακτικής που ακολουθούμε όταν πηγαίνουμε σε διαπραγματεύσεις δια ε, συναπόφασης με στόχο να υπάρξει απόφαση σε επίπεδο πρώτης ανάγνωσης. Νομίζω ότι έτσι μπορείτε να κατανοήσετε αυτό το νέο άρθρο 70α και το επιβεβαιώνει η σωματική γλώσσα της γραμματείας. Λοιπόν, εντάξει, δεν θέλετε περαιτέρω διευκρινήσεις. Ούτως εχόντων των πραγμάτων άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την ε, ομάδα διαπραγμάτευσης και για τον τρόπο διαπραγμάτευσης. Άρχεται. Πέρας. 37 υπέρ, 3 κατά, 2 αποχέ. Σας ευχαριστώ για την εντολή με την οποία με έχετε περιβάλει. Και σας λέω μονάχα ότι εκπλήσωμεν ο λίγων, γιατί σε καμία από τις συζητήσεις που είχαμε είτε στην Ολομέλεια, είτε στην Επιτροπή μας, είτε μεταξύ των σκιωδών, δεν εφάνει ότι ήταν πρόβλημα να έχουμε μια τέτοια ρύθμιση. Εγώ δεν κατάλαβα ότι κάποια πολιτική ομάδα είχε αλλάξει θέση, αλλά τελικά αυτό δεν αλλάζει τίποτα στις διαπραγματεύσεις που θα μπορέσουμε να διενεργήσουμε με το Συμβούλιο και πάντα μαζί με τον εισηγητή της Επιτροπής Μεταφορών. Σας ευχαριστώ και πάμε στο σημείο 24 έκθεση του κυρίου Χιούς, έκθεση πρωτοβουλία, απειλέ εναντίον τη υγεία στο χώρο εργασία λόγω αμοιάντου και προοπτικέ εξάλληψη του υπάρχοντο αμοιάντου στο σύνολό του. Η τροπολογία 27 έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε τη συμβαστική F υπέρ. Κατά. αποχές να κρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές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 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. J υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. K υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε, αν και πιστεύω ότι απορρίφθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 21 ψήφι υπέρ, 16 κατά, εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 90 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της NV14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV13 υπέρ κατα αποχε αποχές εγκρίνεται. NV15 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV11 υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 100 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Θέλετε να επαληθεύσουμε την 101. 102 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. NV3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτω. 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτω. 105. Υπέρ. Κατά. 105. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε για τα 107. Πέρα στις ψηφοφορίες, 24 ψήφοι υπέρ, 19 κατά, εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111, 12, 13, 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. NV9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 101 ε, μάλλον. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχέ. Να επαληθεύσουμε. Επαλήθευση για την 5. Πέρα τη ψηφοφορία. 4 ψήφοι υπέρ, 33 κατά. 5 εποχέ. Έχετε απόλυτο δίκιο Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Υπέρ. Υπέρ τη έκτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται 14. Υπέρ. Κατά. Αποχέ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 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρασε. 40 υπέρ. 2 ψήφοι κατά. Μία αποχή. Συγχαίρουμε τον εισηγητή μας. Si vous avez encore de la force, δεν έχετε ακόμη δυνάμεις. Να περάσουμε στο 25. Έκθεση του συναδέλφου Χάουιτ. Έκθεση πρωτοβουλίας. Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και πορεία προς μια βιώσιμη ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς. compromis Συμβαστική C. Υπέρ. Παρακαλώ. I'm not Κοιτάξτε Ίσως πρέπει να εξηγήσουμε λίγο καλύτερα τα πράγματα όπως έχουν. Πάρα πολύ σιγά λοιπόν να τα κοιτάξουμε αυτά. Οκ. Okay. Συγγνώμη που μίλησα πάρα πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα, <clears throat> είναι σωστός ο κατάλογος. Θέλω λοιπόν να ε, καταγραφούν ευχαριστήσεις μου προς τη γραμματεία γιατί πάρα πολλοί ανησυχούσαν. Θέλω λοιπόν να το καταγράψετε αυτό ευθύ εξ αρχή. Δεύτερον, για να επιταχυνθεί η διαδικασία υπάρχουν προφορικέ ερωτήσει, αλλά περιλαμβάνονται και στον κατάλογο ψηφοφορία και τι έχουμε αυτέ συμφωνήσει με του σκιώδει ηγητέ. Γι' αυτό λοιπόν να ψηφίσουμε τώρα για να κερδίσουμε χρόνο. Αναφέρομαι στις 26 και 1.30 και τέλος, για να ξεπεραστεί το πρόβλημα ότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, παράγραφοι στις ε, γνωμοδοτήσεις άλλων επιτροπών, ε, συμφωνώ με αυτό που είπε η γραμματεία, δηλαδή ότι θα πρέπει να δούμε λιγάκι την ψηφοφορία Υπάρχει λοιπόν μια λογική σειρά και ενδέχεται να πρέπει να υπάρχουν νέες επικεφαλίδες. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και κατά τα άλλα ελπίζω να μην υπάρξουν προβλήματα στη ψηφορία. Ωραία. Κατάλαβα. Η παρέμβαση του εισηγητού δεν έχει καμία, κανένα αντίκτυπο στον κατάλογο των ψηφοφοριών όπως διανεμήθη στις ομάδες. Θα ευχαριστήσω πάντως τους σκιώδεις εισηγητές και όλα τα μέλη της γραμματείας που εργάστηκαν χθες ως αργά για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε σωστά σήμερα το πρωί. Κατάλαβα καλά το πνεύμα της παρέμβασης σας, κύριε Χάουιτ. Ωραία. Εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, ας περάσουμε στην πληροφορία αυτή καθ' αυτή με τρόπο αποτελεσματικό. Παράγραφος 1. Συμβαστική Σ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. D. Υπέρ. Κατά. Αποχέ Εγκρίνεται. Γιούρι 5. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 42. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 43. Για τη 42 να επαληθεύσουμε. Εψήφισαν άπαντες. Εδώ κάνω χάρη στους σοσιαλιστές που δεν ήταν στη θέση τους. Πιστεύω ότι ψήφισαν όλοι. 20 υπέρ, 17 κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Όχι, όχι, συγγνώμη. 43. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Ε. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική AA υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. F υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άφετ 1, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά, Με συγχωρείτε, αλλά ψηφίζουμε. Όχι, όχι, πίπτη, δεν θα έπρεπε να την ψηφίζουμε. Α, ωραία, ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Είναι τα ένα, υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της ΑΘΕΤ 1 θα έπρεπε να ψηφιστεί. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Οπότε επιστρέφουμε στην ΑΘΕΤ 1, στο δεύτερο τμήμα, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αυτό δεν επηρεάζει την ψηφοφορία της ΙΝΤΑ 1, 57 ψηφίστηκε, 58 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική, τι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική G, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, η 65 δεν έγινε αποδεκτή. Όπως μας είπε και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, 66 του κ. Χάουιτ υπέρ. Κατά, αποχές, δεν είναι σαφές, να επαληθεύσουμε. τίκλο. Πέρας. 19 υπέρ, 16 κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 70, Λόπε Φοντανιά υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 71, Σίπελ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική AA καταπίπτει. Ψηφίζουμε τη Γιούρι 4 υπέρ. Γιούρι 4 υπέρ κατά αποχές επίνεται. 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 L'amendement 73 de Madame Η 73 Τη κύρια Λόπ Φοντανιέ. Νόμιζα ότι είχατε αντίρρηση κυρία Μονασάτια, αλλά να την επαληθεύσουμε. Εψήφισα να απαντήσω. Πέρασε. 18 υπέρ, 20 κατά. Σας ευχαριστώ κυρία Σαρτιέ που ζητήσατε την επαλήθευση για την 73 της κυρίας Λόπε Φοντανιέ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα έχει λόξιγκα. 74 και 75. Η κυρία Σάγια. Θα μπορούσατε να δείτε μήπως είναι πλεονάζοντες οι σοσιαλιστές. Νομίζω είναι περάριθμοι. Κάποιος περισσεύει. Έτσι είναι. Πρόεδρος. Όχι. Εάν ήταν ένας παραπάνω οι σοσιαλιστές θα το είχα καταλάβει. Θα το έβλεπα. Και αν δεν το έβλεπα, που μπορεί να συμβεί, θα μου το έλεγε η επικεφαλής τη γραμματείας. Θα το βλέπατε, θα το έβλεπα, γιατί μου το λέει και το μηχάνημα. Θα σα το έλεγα. Καταλαβαίνω όμω και την επαγρύπνησή σα είναι πολύ σημαντική έκθεση για τους σοσιαλιστές 74 και 75. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Δεν εγκρίνεται. Άι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. J υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Amendement 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. και Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκατόν δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. L υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. M υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. N υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Γιούρι 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αφε 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά να επαληθεύσουμε. Άφε 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 34 υπέρ. Μία κατά. Τρεις αποχές. Εγκρίνεται ολοσχερό, αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν τόσο σαφέ. Η ΑΦΕΤ 6 σε δύο τμήματα. Υπέρ, κατά, αποχέ. Να επαληθεύσουμε. ΑΦΕΤ 6. Πέρας. 22 υπέρ, 16 κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα καταπίπτει αυτό. Άφετο 8. Ο εισηγητής είναι κατά υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ. Όχι, αποσύρθηκε 116. 117 υπέρ. Κατά. Από. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές να επαληθεύσουμε για την 117. Εψήφισαν πάντες πέρας. 22 υπέρ. 13 κατά. Εγκρίνεται. Π. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Q. Υπέρ. Για την 118 του Πρέπει να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα, το οποίο είναι προσθήκη στη συμβαστική π. Ποιο είναι υπέρ αυτού του δεύτερου τμήματο, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Να επαληθεύσουμε για το δεύτερο τμήμα, αν και νομίζω ότι εγκρίθηκε. Δεν είμαι βέβαια. Δεν να άπαντε. Πέρασε. 21 υπέρ, 18 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική Q. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 121 υπέρ. 122, 122, συγγνώμη. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 124 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. R υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 129, 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 130 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. S υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΑΦΕΤ 10 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται. 136 υπέρ κατά απόχέ. υπέρ τη 136 υπέρ 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άφετ 15 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κοιτάξτε, προφανώς απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα του της 15. Άθε 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 άφετ. 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Να επαληθεύσουμε. 18. Άφετ 18. Πέρας. 21 ψήφι υπέρ. 17 κατά. Εγκρίνεται. Άφετ 19. Είναι τα 22 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Το ζήτησε η Γκουέ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, και πάλι εγκρίνεται. Άφετ 20 υπέρ. Κατά απόχέ απορρίπτεται. 26, είναι τα 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 147 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά Αποχέ να επαληθεύσουμε για το 152 άρχεται η ψηφοφορία εψήφισαν άπαντες πέρας 23 ψήφοι υπέρ 13 κατά εγκρίνεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε για την 158. Εψήφισαν άπαντες πέρας. 23 ψήφοι υπέρ, 13 κατά, εγκρίνεται. 159 και pour. 159 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 160 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 162 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Με τις ε, επόμενες προφορίες ε, έχω πρόβλημα γιατί δεν ξέρω πώς θα τις πληθήσουμε γιατί η συμβαστική C οδηγεί στην απόρριψη της 164, οπότε περνάμε στην X υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε για την 169. clos. 12. Εψήφισαν άπαντες 12 ψήφοι υπέρ, 18 κατά 9 αποχές. Απορρίπτεται. Ε, 170 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 171 και 172 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Y υπέρ, κατά αποχές Εγκρίνεται. 180 υπέρ. 180 υπέρ. Κατά αποχέ να επαληθεύσουμε για την 180. Πέρα τη ψηφοφορία. 17 υπέρ 22 κατά. Όντω απορρίπτω. 181 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 182 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Z υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 186 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 187 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 188, 189 μάλλον, υπέρ, κατά, Όχι, αποσύρθηκε 188, γι' αυτό ψηφίσουμε τα 189. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε για την 189. Πέρας. 22 υπέρ 17 κατά. Εγκρίνεται. 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. BB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 μάλλον 201 υπέρ. Να ψηφίσουμε για την 202. Όχι, 201. 201 με συγχωρείτε. 201 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Την ψηφίσαμε την ψήση ή κάνω λάθος, όχι, είναι αμέσως μετά. Δεύε 15 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε. Δεύε 15. Πέρα στις προχωριές. 22 υπέρ 17 κατά εγκρίνεται. Συ, συ, συμβαστική σε συ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε 22 κατά πίπτη. ΔΕΒΕ 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άφετε 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν... Μπορούμε να κάνουμε κάτι για τη θέρμανση, είναι σαν να είμαστε στη Σιβηρία. ΔΕΒ 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒ 21 υπέρ, κατά αποχές να επαληθεύσουμε για την 21. Πέρας, 27 υπέρ, 12 κατά, εγκρίνεται. Είναι τα 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Είναι τα 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Είναι τα 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Είναι τα 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Είναι τα 19 υπέρ, κατά, απο, 19, ναι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Είναι τα 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Είναι τα 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα 24 υπέρ. Κατά. Αποχές να επαληθεύσουμε για την ίντα 24. ΙΝΤΑ 24 να πάντες πέρα. 34 υπέρ. 5 κατά. Οπότε πραγματικά ψηφίζεται πανηγυρικά. 36 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κουλτ 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κουλτ 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κουλτ 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μα δεν υπάρχει πρόβλημα να ψηφίσουμε τι 16 και 19, δεν υπάρχουν αντιρρήσει. 16 και 19 μαζί λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτονται. 20 κουλτ. Υπέρ, κατά, να επαληθεύσουμε για την 20. Είναι λιγότερο σαφές. Πέρας. 26 υπέρ, 13 κατά,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 να επαληθεύσουμε για την 9. Πέρα, κύριε Τόμας Μάν, δεν είναι πάντοτε υπέροχο ο κόσμος μας. Έχετε δίκιο, 10 προς 26 δεν εγκρίνεται. Α, 13, υπέρ. Κατά. Υπέρ τη 13. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε και τη συμβαστική B. Την ξέχασα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κύριε Τόμας Μαν, θα το δούμε μετά. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 17 έως 19 τις πληθούσουμε συνολικά υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 21 δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ Πού είναι το αρνητικό. Ε, παρακαλώ να μου τα λέτε εγκαίρως. Μόνο εγώ έχω το λόγο. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 26 ψήφοι υπέρ, 1 κατά 11 αποχές. Συγχαίρουμε τον εισαγητή μας. Και του ευχόμαστε καλές διαπραγματεύσεις με την ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Όχι, νομικών υποθέσεων. Λέγουν ορισμένοι τινές, λέει η πρόεδρος και διακόπτεται. C'était Μήπως μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού την 55 και την 53. και την 55. Όχι, όχι, όχι. Πάλι. Για να είναι σαφή τα πράγματα. Και για τα πρακτικά. Η κυρία Όιμεν Ρόιτεν θέλει να επιταχύνει κάπως τη διαδικασία. Αλλά ίσως δεν γίνεται. Πάμε στην έκθεση του κύριου Μπουλόν για την ε, Ένωση των Υπερποντίων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Overseas Association Decision. Για το σχέδιο αυτογνωμοδότησης προς την Επιτροπή προς την Επιτροπή ΔΕΒΕ Ανάπτυξη ψηφίζουμε από την τροπολογία 52 στην 55 υπέρ κατά αποχές δεκτές συμβαστική αφα υπέρ κατά αποχές δεκτή. 58-25 από κοινού υπέρ κατά αποχές δεκτές. 60 63 όλες μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτές. Συμβαστική β' υπέρ <clears throat> κατά αποχές δεκτή. Μπορούμε να ψηφίσουμε από 65 ως το 41. 65 με 35 υπέρ ψηφίσμα από εκείνου κατά αποχές. 36 υπέρ κατά αποχέ θα ελέγξουμε με ηλεκτρονικά μέσα. Δεν είναι μόνο η κυρία Όμιν Ρόιτον και άλλοι έχουν άλλε απόψει. Πέρα τη προφορία για την 36. 25 υπέρ, 12 κατά, 12 ήταν κατά. Ε, η 36. Είναι σχεδόν ορατή η μειοψηφία αυτή και αναγνωρίσιμη. Δεν θέλουμε να έχουμε διακρίσεις. Λοιπόν, 37 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. 38 με 41 μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού. Εντάξει. Υπέρ. Κατάποχέ εγκρίνονται. 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Όχι. Φωνάζουν. 42 απορρίπτεται. Εννοούσε αυτό. εννοούσα, 43 υπέρ. Κατά αποχές. Αποχές. Απρί, απρίπτεται. Προπολογία 1 υπέρ. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 3 εισηγητής υπέρ κατά αποχές δεκτές. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή 47 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτει 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτει Δελέξουμε 48 Le vote 25, 12 και μία αποχή. 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 49 υπέρ. Κατά αποχές απολύτω. 50 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές αποδεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχέ. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεύτερο τμήμα της 50 κοντά. Πέρας. 20-17 εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 10 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές δεκατή. «51 σε δύο δόσεις. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Το σύνολο της γνωμοδότησης ως έχει τροποποιηθεί. Ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 35-1 με καμία απόχες. Συγχαρητήρια κύριε Μπουλάν που απουσιάζουν είναι. Εγκρίνεται λοιπόν. συνεχαρητήρια Δύο ακόμα μένουσι. Ξέρω ότι έχουν έρθει κάποιοι από τους προσκεκλισμένους μας για την ακρόαση, αλλά σας ζητώ εξ αρχής συγγνώμη. Μπορείτε να γητευτείτε από τη διαδικασία ψηφοφορίας, δεν το κάνουμε επίτηδες, αλλά μπορείτε να την παρακολουθήσετε αν θέλετε. Πρώτο ξεκινήσουμε την ακρόασή μας. Σημείο 27. Η γνωμοδότηση της κυρίας Τσίμερ για τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην ιότητα των ισότητα των φιλοκύρια σήμερα. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα να δώσω μια ένδειξη. Πρόκειται για την τροπολογία 60-61-62. Θέλω να σας υπενθυμίσω εδώ ότι δεν πρέπει να υπάρξει εδώ καμία σύγχυση γιατί πρόκειται για τα συστήματα ελαχίστου εισοδήματος τα οποία διαγράφονται με αυτές τις τροπολογίες. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι πολλές φορές ε, στο παρελθόν επανειλημμένα έχουμε εκφράσει μια θετική άποψη για το ελάχιστο εισόδημα στις εκθέσεις μας. Λοιπόν, εδώ τίθεται ένα αμφιβόλο το σύστημα ελάχιστου ε, εισοδήματος, όχι συστήματα όμως ελαχίστων μισθών. Επομένως δεν πρέπει να υπάρξει καμία σύγχυση. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνέβαλαν στο να υπάρξει αυτή η συμβαστική λύση. Ωραία. Θα ψηφίσουμε με αυτή τη διευκρίνηση συμβαστική α υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική ζ υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική β υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική σε υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μα ψηφίσαμε τη συμβαστική σε. κατά αποχές ενεκρίθη. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική ε υπέρ κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 σε δύο τμήματα. Πρώτη δόση υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Συμβαστική I υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές ή ηλεκτρονικός έλεγχος για την 26 πέρασε 25-13 με 0 αποχές 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή, ακόντα με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμφερτική F υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική J υπέρ αποχές δεκτή. Τροπολογία 42. Υπέρ. Κατά. τη κυρία κυρίας Ροντσούλη, η συγκεκριτή είναι υπέρ. Υπέρ, υπέρ τη 42. Κατά. Αποχέ. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 20, 14 με 4 αποχές γίνεται δεκτή. 43 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 45 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 46 με προφορική τροποποίηση υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 47 τα ίδια υπέρ. Σαν Έχουμε δύο προφορικές τροποποίησεις και ουχή μία να θέτω σε ψηφοφορία τη 47 με τι δύο προφορικές τροποποιήσει υπέρ κατά αποχές δεκτή 48 υπέρ κατά αποχέ δεκτή 50 κοντά υπέρ κατά αποχέ δεκτή 52 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε την 52 Alors, nous vérifions. Ελέγχον, πέρας της ψηφοφορίας. 7 υπέρ δαμία κατά απορρίπτεται. Τι, κλαίρμα. Et donc nous votons le 51. Pour... Ψηφίσουμε την 51 υπέρ. Κατά. Απόχες. Θα λέξουμε και εδώ. Vote clos. 16. με 22. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά αποχέ. Δεκτή. 54 συμβατή υπέρ. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 59 υπέρ κατά έχει δεκτή. Πάλι θα ζητήσω να μας βγάλουν από τα σιβηρικά γκουλάγ σε ό,τι αφορά τη θέρμανση, λέει η πρόεδρος. Είναι ακόμα πιο κρύο τα... 60. Δεν ξέρω τι θέμα έχει στη Λισαβόνα, μήπως πάμε εκεί ή στην Αθήνα. Α, για λόγους αλληλεγγύης. 60 σε δύο τμήματα υπέρ. Κατά. απόχειες απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Εκπίπτει όμως το δεύτερο τμήμα. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα λέξουμε 61. 18 υπέρ, 20 κατά. Ε, από... 62. Στα δύο υπέρ. Κατά. Στα δύο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται 63. υπέρ κατά αποχές απολύτω. 64 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή συμβαστική ντε υπέρ κατά κατά δεκτή 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, δεκτό 68 υπέρ 67 δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικός έλεγχος συζητήθηκε άρχεται η ψηφοφορία πέρας 18 υπέρ 19 όμως κατά δεν γίνεται δεκτή 68 Κυρία Πρόεδρε, για τα πρακτικά θέλω σας πω ότι έκανα λάθος, ψήφισα λάθος, πήγε το χέρι μου αλλού. Θα αναφερθεί στο, στα πρακτικά, αλλά δεν αλλάζει τίποτα αυτό. Μόνο στην Ολομέλη και μετά στις διαπραγματεύσεις μπορεί να υπάρξει κάποια τροποποίηση. 68 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 71 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 72 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότηση ηλεκτρονικά ψηφίζουμε τώρα. Όλοι ψηφίσατε. Πέρασε. 37 1 με 0 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγητρία μας την κυρία Τσιμά. Τελευταία ψηφοφορία της πρωίας, σημείο 28, είναι η έκθεση πρωτοβουλίας της κυρίας Νάντια Ήρσ για την ενσωμάτωση των μεταναστών, τα αποτελέσματα στην αγορά εργασίας και την εξωτερική διάσταση της ε, διαδικασίας συντονισμού των κοινωνικών πολιτικών. Κυρία Μπλίνκεβιτσι, ούτε έχετε το λόγο, εάν το επιθυμείτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να αποσύρω την τροπολογία μου. Η κυρία Μπλικέτσιβούτε αποσύρει την τροπολογία 93 για την παράφο 7. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί έχετε την τροπολογία 92 η οποία είναι μη αποσυρθής εκτός αν κυρία Τζιν Λάμπερτ την αποσύρει. Η κυρία Λάμπερτ την αποσύρει την 92. Τώρα πράγματι οι τροπολογίες 92 αλλά και 93 έχουν αποσυρθεί. Οπότε δεν υπάρχει κανένα αίτημα για διαγραφή του άρθρου 7, της παραγράφου 7. Είναι διάφανη και κρυστάλλινη σε σαφήνεια η κατάσταση. Πάμε στη ψηφοφορία λοιπόν. Σύμβαστη, J. Υπέρ. Δεκτή. Λίμπε 2. Υπέρ κατά. Λοιπόν, νομίζω μπορούμε να ψηφίσουμε την παράγραφο 2 της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, η οποία είναι ως προστίκη. ΛΥΜΠΕ 2 υπέρ κατά αποχές υπέρ. Δεκτή. Λίπε 7 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Συμβαστική S υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική K υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 51 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Φεμ 20 υπέρ. Κατά αποχές. Θα ελέγξουμε. πέρασε. 17, δεν εγκρίνεται. 25 φαμ υπέρ κατά αποχές. Δεν βλέπω να ψηφίζει κανείς. 25 πάλι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Παρακαλώ να παρακολουθείτε. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές δεκτή. 56 και αποσυρθεί. Η ε, e, υπέρ δεκτή. Λίμπε 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΦΑΜ 12 υπέρ κατά αποχές. Θα έλεξουμε. 14 14-17 δεν γίνεται δεκτή. Φαμ 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική εμ υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 63 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική εν υπέρ κατά αποχές δεκτή. 71 Χίρς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ο υπέρ Έλεγχος για την 71, εντάξει, άρχεται. Αφού απορρίφθηκε όμως γιατί την ελέγχουμε. Πέρασε στις προφορίες. 6.28 με, με μία αποχή. Οι φιλελεύθεροι οι οποίοι είναι επάγρυπνοι και οξυδερκείς γιατί δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Γιατί δεν εώρακαν αυτό το οποίο έλαβε χώρα στην 71. Απερίφθη λοιπόν. Συμβαστική ο, υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική υπέρ, υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΦΑΜ 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΦΑΜ 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΦΑΜ 3 υπέρ Si monsieur, si monsieur Horry se trompe là, je suis perdu. Donc vous voulez... Έκανε λάθος ο κύριος Horry. Αλλά... Τέλεχος στην 11 γυναικών. Ωραία, πάμε. On vérifie le Le vote est clos. 18, 17. Γίνεται δεκτή. Γίνεται δεκτή. Τρία γυναικών υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική R υπέρ κατά αποχές δεκτή. Κομπρομητή και πούρ. Βαστείτε, τε, κατά αποχές, δεκτή. Συγγνώμη. 95 υπέρ. Κατά αποχές θα ελέγξουμε την 95. Πέρασε. 23-12 εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ου υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ε, κατά 100 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική δε υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική τροπολογία W υπέρ κατά αποχές δεκτή. 26 φαμ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 107 κοστέλο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 108. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποδεκτή. 19 λίμπε. Υπέρ κατά αποχές δεκτή, 24 λίμπε υπέρ κατά αποχές δεκτή. 118 υπέρ κατά χέσα. θα ελέγξουμε την 118 πέρας 10-22 απορρίπτεται συμβαστική ε, Y υπέρ κατά αδεκτή συμβαστική Z κατά αποχές δεκτή 131 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 132 υπέρ. Κατά. Γιατί δεν ψηφίζετε, γιατί, γιατί, 132 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική, α, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική, μπιμπι, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 147 υπέρ κατά αποχές δεκτή 153 υπέρ κατά αποχές δεκτή 154 υπέρ κατά αποχές δεκτή 155 υπέρ κατά αποχές δεκτή 156 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Κατά υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 3 αφέτ υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 163 ή τι εισηγήτριες υπέρ κατά αποχές δεκτή. 164 Λάμπερτ υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αφέτ 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 165 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική σε υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 φαμ υπέρ κατά 27 φαμ υπέρ κατά αποχές δεκτή 169 υπέρ κατά αποχές δεκτή απορρίπτεται 170. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 171. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Αφέτ 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Αφέτ 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 173 ότι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστή ΔΕΝΤΕ. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 172 δεν είναι δεκτή. Λίμπε 12 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Λίμπε 10 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Φαμ 19 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Φαμ 9 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 179 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Φαμ 15 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστή ΕΕ υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική FF υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική GG υπέρ κατά αποχές δεκτή. 188 υπέρ κατά δεκτή. 189 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 190 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Απολύπτεται. 191 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Θα έλεξουμε την 191. Δεκτεί, δεκτεί, δεκτεί, δεκτεί, μην ελέγχεται. 193 και 94 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 195 υπέρ, κατά αποχές υπέρ, 195. Αποχές δεκτή. Ας, ας, έτσι, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 197 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 199 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Φάμ 22 υπέρ κατά αποχή δεκτή. Φάμ 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ερχόμαστε αιτιολογικές αναφορές. Τροπολογία 1 υπέρ κατά δεκτή. Όλες μαζί. Α, όλες με. 1 με 8 όλες μαζί υπέρ κατά αποχές δεκατές. 10 υπέρ <clears throat> κατά αποχές δεκτή. Αιτιολογικές σκέψεις. 11 όντι υπέρ κατά αποχές δεκτή. ένα λιμπέ υπέρ κατά αποχές δεκτή. δώδεκα καμπρονιό υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική β υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική σε υπέρ κατά αποχές δεκτή. Φαμ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φαμ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 ότι υπέρ κατά. Θα ελέγξουμε την FAM G. G FAM. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Καταλάβατε. 33 με μία κατά ψήφο μονάχα. 19 ότι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 Στάινοκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστή Ντε υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΣΕ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΜΠΕ υπέρ κατά Φαμπέ υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές δεκτή. 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές δεκτή. 35 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές δεκτή, 36 υπέρ κατά αποχές δεκτεί. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 θα ελέγξουμε. Πέρασε. 17-17 απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική ή e, τελευταία, τελευταία υπέρ κατά αποχές δεκτή, γίνεται δεκτή το σύνολο της ε, έκθεσης με την τελευταία ηλεκτρονική ψηφοφορία της ημέρας άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Α, βγάλατε πολύ γρήγορα τις κάρτες σας. Όχι, όχι, κρατήστε τις κάρτες σας μέσα. Δεν τελείωσε ακόμα. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάμε. Πάμε. Ωραία. 34-0. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μείνατε στο τέλο. Παλικάρια. Συγχαρητήρια στην κυρία Χέρι. Ομόφωνα δεκτή η έκθεσή τη. Σουτ. Όσοι θέλουν να φύγουν να το κάνουν σιωπηρός. Έχουμε καθυστερήσει για το επόμενο σημείο που είναι πολύ σημαντικό είναι στα πλαίσια της έκθεσης Lambert το σημείο 30 δημόσια κρόαση για τα αποτελέσματα της κρίσης σε σχέση με την πρόσβαση σε περίθαλψη για τις ευάλωτες ομάδες. 30 δευτερόλεπτα διακοπή της συνεδρίας. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην Jean Lambert για να κάνει μια εισαγωγή στην ε, ακρόαση και μετά θα δώσω το λόγο στους εισηγητές. Θέλω να τους ευχαριστήσω και τους τέσσερις. Αλλά σας πενθυμίζω ότι η εισηγήτρια λαμβάνει το λόγο για να θέσει το πλαίσιο των επικειμένων παρεμβάσεων. Έχετε το λόγο Jean Lambert. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και αυτούς οι οποίοι είναι παρόντες σήμερα. Υπήρχαν και άλλοι φορείς οι οποίοι ήθελαν να λάβουν το λόγο μαζί μας για τα θέματα αυτά, για την πρόσβαση στην περίθαλψη. Πολλοί από εμά ενετυπωσιάστηκαν από ορισμένε εκθέσει κάτι κράτη-μέλη σε σχέση με άτομα τα οποία δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διάφορες μορφές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λόγω κόστους κτλ. Και νομίζω ότι γνωρίζουμε ότι η δημόσια υγεία δεν είναι αρμόδια, δεν αρμοδιότητα της Επιτροπής μας, αλλά προφανώς ο κοινωνικός αντίκτυπος έλλειψης περίθαλψης είναι θέμα δικό μας. Χθε στην προφορική ερώτηση που υποβάλαμε με το Ευρωπαϊκό, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανεξάρτητη Διαβίωση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν περαιτέρω πιέσεις στους ε, απλούς ανθρώπους που έχουν όλο και περισσότερες δυσκολίες να έχουν μια αυτονομία και μια ζωή αξιοπρέπεια λόγω της κρίσης. Αυτό λοιπόν που θέλαμε να δούμε σήμερα είναι πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα κατά τη διάρκεια της κρίσης για ορισμένες ευάλωτες ομάδες. Δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ομάδες ποια είναι η άποψη των ανθρώπων αυτών που πλήττονται για τα συστημικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αν υπάρχουν προτάσεις για να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε τα θέματα αυτά. Η Κομισιό μιλάει για προγράμματα κοινωνικής καινοτομία. Θα βοηθήσει βέβαια κανένα αυτό το πράγμα ή θα πρέπει να εξετάσουμε άλλες προσεγγίσεις για τα άτομα αυτά τα οποία χρειάζονται να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην περίθαλψη, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι παιδιά, είτε είναι άτομα με αναπηρίες, προβλήματα με ιδιαίτερε ιατρικές ανάγκες που είναι ήδη ευάλωτα, οι φορείς HIV, AIDS κτλ. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διατυπώσουμε προτάσεις, καταρχήν να εντοπίσουμε ποια είναι τα προβλήματα και να καταθέσουμε προτάσεις για την αντιμετώπιση του. Είμαι λοιπόν πολύ ευγνώμων για την παρουσία όλων των ομιλητών σήμερα και όπως ξέρετε είναι και άλλες ομάδες που μα έχουν δώσει γραπτά πληροφορίες σε μένα την ίδια και φυσικά την κρατώ την πληροφορία αυτή στη διάθεση όλων αυτών που θα θέλαν να ξέρουν κάτι περισσότερο. Ε, ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον Νικήτα Κανάκη, εξ ονόματος των γιατρών του κόσμου και θέλω να χαιρετήσω την παρουσία μιας αντιπροσωπείας από το Νομαρχιακό Συμβούλιο των Πυρηνέ Ατλαντικ με τον Ζωζ Επικεφαλή. επικεφαλής. Καλώς ήλθατε στις Βρυξέλλες για να παρουσιάσετε τα επιχειρηματά σας και είμαστε πράγματι έτοιμοι να σας ακούσουμε. Είτε στα πλαίσια του ΦΕΝΤΕΡ είτε του Κοινωνικού Ταμείου. Ο λόγος τώρα στον κύριο Νικητά Κανάκη, εξ ονόματος των ιατρών του κόσμου. Κυρία Πρόεδρε, Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Ehre, die Sie uns erweisen, dass wir heute hier sein dürfen. Αναφορικά με τις επιπτώσεις της κρίσης στη δημόσια υγεία και στην πρόσβαση των ανθρώπων. Έχουμε καταθέσει και έχετε ένα πλήρες κείμενο που αναφέρει πολλές από τις απόψεις μας, πολλά από αυτά που υποστηρίζουμε και αυτά που προτείνουμε. Θα προσπαθήσω μέσα σε ελάχιστα λεπτά να σας δώσω μια εικόνα δίνοντας έμφαση στο παράδειγμα της Ελλάδας από όπου προέρχομαι, μια και στο δίκτυο των γιατρών του κόσμου θεωρούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μια εξαίρεση στην κοινή πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένα παράδειγμα το τι μπορεί να συμβεί όταν η οικονομική κρίση αγγίζει τους ανθρώπους. Σήμερα το δίκτυο των γιατρών του κόσμου αντιπροσωπεύει 15 χώρες με περισσότερα πέρα από τη δουλειά εκτός Ευρώπης, 324 εθνικά προγράμματα που προσπαθούν να υπηρετήσουν μια πολύ απλή αλήθεια που για μας είναι η βάση της ιατρικής ηθικής. Ότι το δικαίωμα, η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη είναι δικαίωμα και δεν είναι πολυτέλεια. Αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε για τους πιο φτωχούς από τους ανθρώπους που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε είναι μετανάστες, είτε είναι άνθρωποι που ζουν στο δρόμο, είτε είναι τσιγκάνοι, είτε είναι ανασφάλιστοι που συναντάμε όλο και περισσότερο. Μια πρώτη, αν θέλετε, σημείωση έχει να κάνει ότι αυτό που ζούμε κυρίως στον Νότο με την οικονομική κρίση δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο να οδηγήσει σε μια μεγάλη κοινωνική αποσάρθρωση. Δεν είναι απλά μόνο το δικαίωμα στην υγεία το οποίο μειώνεται καθημερινά, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι σε χώρες όπως για παράδειγμα η Ισπανία όπου ήταν ένα πρότυπο καλής πρακτικής ενσωμάτωσης σήμερα καλούνται οι γιατροί να απομακρύνουν ουσιαστικά από τα νοσοκομεία αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο είναι ένα πρόβλημα που οδηγεί πολλούς πολίτες και ανάμεσά τους αναφέρομαι κυρίως στην Ελλάδα να αισθάνονται ότι μέσα στην ίδια την Ευρώπη που είναι μέλη είναι αποκλεισμένοι. Απευθύνομαι περισσότερο στο συναισθημά σας, διότι γνωρίζω ότι μοιράζεστε αυτές τις αγωνίες με τους πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών που σας έχουν εκλέξει εδώ. Και αναφέρω ότι οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι στην Ελλάδα σήμερα βρίσκονται σε μια πάρα πολύ μεγάλη δύσκολη θέση. Τα στοιχεία τα οποία θα έχετε στη διάθεσή σας στο κείμενο που, που σας έχουμε καταθέσει δείχνουν ότι στα ιατρία των γιατρών του κόσμου που δίνουν δωρεάν ιατρική φροντίδα σε όσους δεν συμμετέχουν στο σύστημα υγείας και αποκλείονται έχουν, έχει εξαπλασιαστεί ο αριθμός των Ελλήνων πολιτών από το 10% σήμερα στους περίπου 40.000 ασθενείς που σε όλη την Ελλάδα έρχονται ζητώντας δωρεάν ιατρική φροντίδα έχει ανεβεί στον αριθμό του 50%. Σε μερικά δε ιατρία περιφερειακά έχει ξεπεράσει το 80% και το 90%. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μέχρι πριν 2-3 χρόνια είχαν μια κανονική ζωή. Ήταν άνθρωποι που ήταν πλήρως ασφαλισμένοι και που ξαφνικά νιώθουν ότι βρίσκονται εκτός. Θυμίζω για όσους πιθανόν δεν το γνωρίζουν ότι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, αν είσαι άνεργος μετά από ένα χρόνο, δεν έχεις ούτε εσύ ούτε η οικογένειά σου κανένα απολύτως ασφαλιστικό δικαίωμα, με αποτέλεσμα να μην μπορείς να φτάσεις ούτε στα βασικά στο σύστημα υγείας, που έτσι κι αλλιώς πια απαιτεί ένα εισιτήριο σήμερα 5 ευρώ και σύμφωνα με τις επιταγές της Τρόικα τη χρονιά που έρχεται 25 ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση μεταναστών. Σας μεταφέρω εδώ περισσότερο από τα νούμερα την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Την αγωνία των γονιών που βλέπουν στα πολυετρία να έρχονται των γιατρών του κόσμου για να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, διότι τα παιδιά αυτά δεν δικαιούνται εμβολιασμό, παρόλο που είναι Έλληνες πολίτες. Και το είναι ό,τι πιο άδικο μπορεί να συμβεί σε αυτά τα παιδιά. Σας λέω μόνο ότι μόνο φέτος έχουμε εμβολιάσει περισσότερο από 8.000 παιδιά, 8.000 δηλαδή οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν, άρα υπήρχε και ένα σοβαρό πρόβλημα πρόσβασης λόγω του μη εμβολιασμού στην εκπαίδευση. Σας μεταφέρω την αγωνία ηλικιωμένων ανθρώπων οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ζουν με εισοδήματα όπως προκύπτει από τα στοιχεία μας με λιγότερα από 300 ευρώ το μήνα σε μια χώρα που είναι σχετικά ακριβή και οι οποίοι δυσκολεύονται να βρούνε τα φαρμακά τους. Όποιος έχει μια χρόνια πάθηση όπως για παράδειγμα διαβήτη ή μια καρδιοπάθεια η καθημερινή επιβίωση γίνεται γι' αυτόν γολγοθάς. Σας μεταφέρω την αγωνία εγγύων γυναικών οι οποίες επειδή είναι ανασφάλιστες δεν έχουν το δικαίωμα στη δωρεάν φροντίδα και στη δωρεάν, στο δωρεάν τοκετό, καλούμενοι πολλές φορές να πληρώσουν χρήματα τα οποία δεν έχουν. Σήμερα... Θα μιλήσω συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, μου είπαν ότι ο μεταφραστής ε, δυσκολεύεται. Ζητώ συγγνώμη που μιλάω γρήγορα, αλλά δεν έχω συνηθίσει να βρίσκομαι και θα προσπαθήσω να μιλήσω λίγο πιο αργά. Ε, θα σας μεταφέρω επίσης την αγωνία ανθρώπων οι οποίοι πλέον δεν βρίσκουν τρόφιμα, δεν βρίσκουν ούτε τα βασικά τρόφιμα και έρχονται αναζητώντας ακόμα και τα πιο απλά πράγματα. Θυμίζω ότι το ελληνικό κράτος ήδη έχει ξεκινήσει να δίνει συσίτια στα σχολεία, άρα ξαναγυρίζοντας σε εποχές πολλών δεκαετιών πίσω. Τι προσπαθώ να πω με όλα αυτά. Προσπαθώ να ισχυριστώ ότι η έλλειψη πρόσβαση στο σύστημα υγείας για τους πιο φτωχούς οδηγεί σε κοινωνικά προβλήματα τα οποία πολύ σύντομα θα είναι απρόβλεπτα. Θυμίζω, γιατί το ζούμε και αυτό στα ιατρία των γιατρών του κόσμου, σε όλη την Ευρώπη αλλά κυρίως στην Ελλάδα, ότι έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η ξενοφοβία, ο ρατσισμός. Συναντάμε ακραίες ομάδες να συναντούν όλο και μεγαλύτερη λαϊκή αποδοχή, κυρίως λόγω του θυμού του κόσμου ο οποίος αποκλείεται. Έρχομαι λοιπόν και ισχυρίζομαι εκ μέρους όλου του δικτύου ότι πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή την πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Ισχυριζόμαστε και νομίζω ότι αποδεικνύεται στα κείμενα τα οποία έχουμε καταθέσει ότι η, έλλειψη πρόσβασης πιθανότατα θα κοστίζει πολύ περισσότερο από το όποιο κόστος θα είχε η πρόσβαση ε, ανθρώπων που σήμερα αποκλείονται. Ακόμα και για όσους αγαπούν τα νούμερα, εγώ δεν τα πηγαίνω πολύ καλά γιατί είμαι γιατρός, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι η μη η μη πρόσβαση, το να μην λύσει ένα πρόβλημα μπορεί μακροχρόνια να σου κοστίσει πολύ περισσότερο, χωρί βεβαίω να αναλογιστεί κανένα τι συμβαίνει με τα θέματα δημόσια υγεία. Τέλο, και θα σταματήσω εδώ, δεν θέλω να καταχραστώ άλλο το, χώρο, το χρόνο. Πρέπει να θυμίσω, να, να, να φέρω επίσης ε, υπόψη σας μια καινούργια πραγματικότητα την οποία μέχρι πριν λίγο καιρό αγνοούσαμε. Η οικονομική κρίση οδηγεί όλο και περισσότερου ανθρώπου να μετακινούνται εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαίου πολίτε αναζητώντα δουλειά και καλύτερε μέρε σε άλλε χώρε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ανασφάλιστοι. Αυτοί οι άνθρωποι δυσκολεύονται σε όλη την Ευρώπη όλο και περισσότερο να βρούνε πρόσβαση στα συστήματα υγείας. Δεν είναι μόνο Έλληνες, είναι Ισπανοί, είναι Πορτογάλοι, είναι άνθρωποι από τη Βουλγαρία ή από τη Ρουμανία. Είναι ένα καινούριο πρόβλημα το οποίο πρέπει να το δούμε διότι δημιουργεί φραγμούς και στην ελεύθερη μετακίνηση αλλά πολύ περισσότερο δεν δίνει τη δυνατότητα στου πιο φτωχού ανθρώπου που αναζητούν μια καλύτερη μοίρα να είναι υγιεί ώστε να έχουν μια καλύτερη πρόσβαση στην υγεία. Τέλος, θέλω να επισημάνω και θα σταματήσω με αυτό, την πάγια διεκδίκηση των γιατρών του κόσμου, όταν αφορά μετανάστες, ανθρώπους άσχετα αν έχουν ή δεν έχουν διοικητικά χαρτιά, αλλά κυρίω αυτού που δεν έχουν, που καταφεύγουν οικέτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν σοβαρά προβλήματα υγεία, να μην απελάβνονται, να μην επιστρέφουν στι χώρε του, να μπορέσουμε να του δώσουμε έστω και στοιχειώδη φροντίδα, όχι μόνο γιατί αυτό είναι ηθικό και σχετίζεται με τι ίδιε τι αρχέ τη Ευρώπη, αλλά πολύ περισσότερο γιατί είναι ένα μήνυμα, αν θέλετε, ότι η Ευρώπη συνεχίζει να είναι αυτό που εσείς υπηρετείτε και όλοι θέλουμε ένας χώρος καταρχήν κοινωνικής αλληλεγγύης, δημοκρατίας, βασισμένος στις πιο σημαντικές από τις ευρωπαϊκές αξίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Euh, ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα στο δεύτερο παρεμβάνω, παρεμβάνω στον Μισελ Λεγκρό, αλλά θέλω να χρησιμοποιήσω το άρθρο 9 του κανονισμού Ο Ζομπερές ήταν συνειδητής των ε, ιατρών του κόσμου, θα ήθελα αυτό να το αναφέρω και δίνω το λόγο στον Μισελ Λεγκρό, ο οποίος είναι υπεύθυνο για τα θέματα ε, δημόσιας υγείας στην Σχολή Υψηλών Σπουδών και μέλος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Ένδια και την κοινωνική, κοινωνικό αποκλεισμό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πέραν των καθηκόντων που αναφέρατε και ίσως αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι και σήμερα μαζί σας, έχω αναλάβει τη Διεύθυνση Υγεία και Πρόσβαση στην Υγειονομική Περίθαλψη που θα ετοιμάζει την εθνική μας διάσκεψη κατά της φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ε, έγινε πρόσφατα τον Οκτώβριο, στις αρχές Οκτωβρίου στο Παρίσι. Ε, κάναμε ένα, μια παρουσίαση πενταετούς προγράμματος, ε, το οποίο εγκρίθηκε και παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό μας την περασμένη Δευτέρα. Αυτά εισαγωγικά. Όταν μιλάμε για κρίση στη Γαλλία και στον τομέα της υγείας αυτή τη στιγμή, περισσότερο αναφερόμαστε σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον αμίαντο, με την αντισύλληψη με την γρήπη, την επιδημία γρήπης ή τις, τα εμφυτεύματα στο στήθος, τα εμφυτεύματα σε λιγόνης. Όμως όχι, οι κριση στην υγεία, στο τμήμα, στο, στον τομέα υγείας είναι περισσότερο θέμα επαγρύπνησης παρά οικονομικής κρίσης. Αυτή είναι μια πρώτη παρατήρηση που πρέπει να έχουμε κατά νου. Ε, έπειτα έχω πολλέ παρατηρήσει να κάνω και να δώσω και κάποιε ιδέε. Πρώτη, διαπίστωση. Όταν αναλύει κανεί το γαλλικό σύστημα υγεία ε, και το, το τοποθετεί στο πλαίσιο τη κρίση, βλέπει ότι δεν υπάρχει ακόμη διακοπή ως προς την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών ή της πρόσβασης στην υγεία των διαφορών ομάδων του πληθυσμού. Ακόμη δεν βρισκόμαστε στην κατάσταση που περιέγραφε ο Έλληνα συνάδελφο ή Ισπανοί συνάδελφοι ενδεχομένω. Δεν υπάρχει κατάρρευση, δεν υπάρχουν κραδασμοί. Αντιθέτω, υπάρχει κάτι άλλο και θα ξανάρθω σε αυτό. Η παράταση των πιέσεων, των εντάσεων που ήδη γνωρίζαμε από κάποια χρόνια στο γαλλικό σύστημα υγεία. Δεν υπάρχει επίση κατανομή του πληθυσμού ή πρόβλημα αποκλεισμό του πληθυσμού που δεν έχει πλέον πρόσβαση στην υγεία ή στι οικονομικέ υπηρεσίε. η στι οικονομικε υπηρεσιε μια κατάσταση που να δείχνει ότι εμφανίζονται νέες παθολογίες. Ε, βεβαίως ε, υπάρχουν κάποια κρούσματα θυματίωσης, κάποιες ε, παθολογίες είναι περισσότερο συχνές σε κάποια τμήματα του πληθυσμού, αλλά παραμένουμε σε καταστάσεις περιθωριακές, περιορισμένες. Δεν θα τα αναπτύξω αυτά τώρα αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα σύστημα υγείας με πολύ υψηλό κόστος, 12% του ΑΕΠ για την υγεία, τρίτη θέση, ε, μετά τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Ολλανδία. Το σύστημά μας επίσης έχει ιδιαίτερα κοινωνικό χαρακτήρα με την κοινωνική πρόνοια και εδώ και 15 χρόνια για τον πληθυσμό με χαμηλό εισόδημα και πέρα της κοινωνικής ασφάλισης έχουμε προβλέψει πρόσθετο επίδομα της ε, καθολικής υγειονομικής περίθαλψης που επιτρέπει το να αποζημιώνονται κάποια έξοδα, ιδίως για όσους είναι μειονεκτούντες. Δεν υπάρχει λοιπόν κατάρρευση. Αντιθέτως, υπάρχει μια επίταση του φαινομένου που θα το ονόμαζα ένα, σύστημα, ένα φαινομένο ψαλίδας, κάτι που έχει παρουσιαστεί εδώ και κάποια χρόνια στο γαλλικό σύστημα. Ε, αυτό είναι ένα φαινόμενο διτό. Από τη μια όπως παντού έχουμε αύξηση της φτώχειας, 14% του γαλλικού πληθυσμού κάτω από το κατόφλι της φτώχειας πλέον. Θυμίζω ότι το κατόφλι της φτώχειας ε, ε, είναι 1900 ευρώ για έναν άνθρωπο που ζει μόνος του. Και επίσης, όπως οι περισσότερες χώρες γνωρίζουμε και γύρανση του πληθυσμού. Από δημογραφικής άποψης, 15% του πληθυσμού ε, που φέρουν από χρόνιες παθήσεις καρδιοαγκιακές, ε, διαβήτη, ψυχιατρικές ε, νόσους και ούτω καθεξής. Επίσης, σε αυτό το φαινόμενο της ψαλίδας έχουμε όλο και περισσότερους μετανάστες χωρίς επίσημα έγγραφα που όλο και πιο δύσκολα έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Πέραν αυτού, η δεύτερη άκρη της ψαλίδας που δημιουργεί αυτό το χάσμα, αυτή τη μεγάλη απόσταση, έχει να κάνει με το ότι προσπαθήσαμε να ρυθμίσουμε και να μειώσουμε τις δαπάνες της υγείας. Το ε, ετήσιο έλλειμμα του συστήματος υγείας στην ε, Γαλλία φτάνει τα 10 δις ευρώ και αυτό προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε. Υπάρχουν προγράμματα διόρθωσης κάθε δύο χρόνια με νέες αποζημιώσεις, με λιγότερες ιατρικές δαπάνες. Επίσης το σύστημα προστασίας στα σχολεία έχει αλλάξει, δεν είναι πλέον τόσο αποτελεσματικό όσο στην αρχή και το ίδιο με την εργασιακή, ε, την ε, ιατρική, προσφορά ιατρικής περίθαλψης στα σχολεία, στην, στην δουλειά, στην εργασία, το ίδιο και στην Ήπεθρο. Ε, Ακόμα και για τους ηλικιωμένους υπάρχει ένα επίδομα που μελετάτε εδώ και κάποια χρόνια. Υπάρχει λοιπόν μια απόσταση που ολοένα και μεγαλώνει. Η κρίση έχει οξύνει την κατάσταση αυτή. Δηλαδή από τη μια έχουμε ένα σύστημα υγείας που αντιμετωπίζει τους οικονομικούς κρατασμούς και από την άλλη μια ένα πληθυσμό που φτωχαίνει και ολοένα γίνεται φτωχότερος. Ε, είναι πιο πολύ άριθμοι οι φτωχοί ε, πολίτες. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με πληθυσμό με χαμηλά εισοδήματα, με λιγότερο καλή κατάσταση υγεία από το γενικό πληθυσμό και με πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη που όλο ένα και δυσκολεύεται, δυσχεραίνεται. Αυτό λοιπόν μας απασχολεί από την άποψη των υπηρεσιών που προσφέρονται σε επίπεδο οδοντιατρικής ή οφθαλμιατρικής βλέπουμε ότι οι πλέον φτωχοί δεν έχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Ένα 17% δεν τις αποζητούν καν, ενώ στον γενικό πληθυσμό με μεγαλύτερα εισοδήματα φτάνει το 17%. Έτσι αυξάνονται οι ανισότητες, προφανώς λόγω των εισοδημάτων, αλλά κυρίως και λόγω της, ε, των περιοχών του γεωγραφικής κατανομής. Υπάρχουν ε, γεωγραφικές περιοχές που είναι ε, περισσότερο φτωχέ με δυσκολότερη πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Υπάρχουν λοιπόν ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού που είναι εκτεθειμένα σε μεγαλύτερους κινδύνους. άνεργοι, εργαζόμενοι με συμβάσεις πολύ συντομιδιακές που δεν μπορούν να έχουν συμπληρωματική ασφάλιση, άνθρωποι που καθυστερούν, αναβάλουν την ε, πρόσβασή τους στο σύστημα υγείας, την ε, παροχή, την λήψη ιατρικών υπηρεσιών, οπότε η κατάστασή τους επιδεινώνεται. Δεν πάνε εύκολα στα νοσοκομεία, στα επίγοντα. Βεβαίω είναι δωρεάν η περίθαλψη αυτή, όμω αντιστρόφω δεν υπάρχει και πρόληψη. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί μόνο όταν υπάρχει επίγουσα ανάγκη θα καταφύγουν σε νοσοκομιακή περίθαλψη. Επίση αυξάνεται ο πληθυσμό όσων δεν έχουν έγγραφα, των μεταναστών δηλαδή επίσημα έγγραφα, και στην Ήπεθρο ε, η κατανομή ηλικιωμένων νέων δημιουργεί μια κατάσταση οξυμένη η ηλικία, και εδώ θα συμφωνήσω με τον Έλληνα συνάδελφο, σε δύο γαλλικέ περιοχές, από τη μια την Μαγιότ, στον Ινδικό ωκεανό και στη Γουιάννα, εκεί βλέπουμε η κατάσταση να είναι ιδιαίτερα δυσχερή. Ταυτόχρονα, αυτό το έχει επιτείνει η κρίση, ε, βλέπουμε ότι η γαλλική κυβέρνηση αποφασίζει κάποια σειρά μέτρων που θα θεσπιστούν, θα ληφθούν. Πρώτη ιδέα, ε, ο χώρος της πολιτικής δεν έχει στοχεύσει τους πληθυσμούς που είναι πλέον μειονεκτούντες, αλλά περισσότερο επανεπιβεβαιώνει την ε, ανάγκη να καταπολεμηθούν οι ανισότητες στον τομέα της υγείας τα τελευταία δέκα χρόνια. Δεν έχουν γίνει στοχευμένες δράσεις, δεν έχουν αναλυφθεί στοχευμένες δράσεις. Αυτές έχουν συμπεριληφθεί σε μια ευρύτερη πολιτική καταπολέμησης των ανισοτήτων δεύτερος άξονας πολιτικής δράσης ήταν η μείωση των ε, ιατρικών ε, δαπανών για τους πλέον ευάλωτους, αυξάνοντας το κατόφλι κάλυψης ε, με, την οικονομική, με το οικονομικό κριτήριο, 700.000 άτομα αφορά περίπου αυτό το μέτρο. Επίσης υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση σε άτομα που δεν χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που τους δίνονται, την οικονομική περίθαλψη, διότι ε, κάποιες φορές ε, αυτό μπορεί να είναι λόγω στιγματισμού από ένα 10 έως 24% αφορά η ομάδα αυτή του πληθυσμού και έπειτα για κάποιες βασικές υπηρεσίες προσφέρονται πιο εύκολα στους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς ώστε να τους προσελκύσουμε στις βασικές υπηρεσίες υγείας. Τελευταία παρατήρηση. Ρόλο τη Ευρώπης. Εδώ να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ιδιαίτερα παρούσα στον χώρο της υγείας στη Γαλλία. Περισσότερο ενθαρρύνει τη μείωση των ελλημάτων λόγω της ασφάλισης παρά την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Η Ευρώπη όμως ε, θα είχε πολλά να ωφεληθεί αν έδινε μεγαλύτερη έμφαση στη μακροχρόνια περίθαλψη, στην πρόληψη και αν συμπεριλάμβανε στην πολιτική ατζέντα θέματα κάλυψης ηλικιωμένων ομάδων του πληθυσμού ή αν έθετε ερωτήματα για την κατάσταση των μεταναστών και όσων δεν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα. Το θέμα αυτό ανακύπτει και σε άλλες χώρες, αλλά και στη Γαλλία. Και έπειτα Ακούγοντα τον Έλληνα συνάδελφο, πρέπει και εγώ να σχολιάσω, επειδή γνωρίζω τι συμβαίνει στι χώρε του Νότου. Προφανώ θα πρέπει να υπάρξει διοργάνωση τη αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδίω σε θέματα υγεία. Δεν θα πρέπει αυτό να παραμείνει θεωρητικό, αλλά να το σχεδιάσουμε και να το υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για αυτήν την μαρτυρία από την Γαλλία που έχει και γαλλική εμβέλεια βέβαια. τρίτο προσκεκλημένος ο κύριος Λουκ Ζέλντελο, Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρεχόντων υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την πρόσκληση που μου απευθύνατε και για το γεγονός ότι μου επιτρέπετε να μοιραστώ μαζί σα τι ανησυχίε μου και κάποια στοιχεία που θέλω να σα παραθέσω σε σχέση με τον αντίκτυπο τη κρίση στο δικό μα τομέα. Νομίζω ότι η έκθεσή μα σα έχει δοθεί σε επίπεδο PowerPoint και θα σας βοηθήσει να παρακολουθήσετε την παρέμβασή Φυσικά, οι κοινωνικέ υπηρεσίε είναι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στον τομέα αυτό γιατί αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή ουσιαστικά υποσκάπτει την ε, εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και των συνδεωμένων μέτρων. Το δυναμικό του κοινωνικού τομέα δεν χρησιμοποιείται σε αυτή τη φάση. Υπάρχουν περικοπές οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα ευθύς και αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα δεν έχει καθόλου περιεκτικό χαρακτήρα. Στα 10 λεπτά που έχω θα ήθελα να τα χρησιμοποιήσω για να σας δώσω ορισμένα στοιχεία επί τη βάση των ερευνών που έχουν γίνει από τον φορέα μου, το ESPD. Θέλω να αναφερθώ όμως και στο υλικό το οποίο μας δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Foundation. Αυτό είναι ένα έγγραφο το οποίο θα δείτε και στην είσοδο σε σχέση με τον αντίκτυπο της κρίσης για τις ευάλωτες ομάδες. Ας δούμε καταρχήν τον αντίκτυπο της κρίσης σε υποστηρικτικού χαρακτήρα υπηρεσίες. Παρακολουθήσαμε την κατάσταση αυτή από το 2009 μέχρι σήμερα και βλέπουμε ότι υπάρχουν τρία αλληλένδετα στοιχεία αντικτύπου. Καταρχήν για τη βιωσιμότητα του τομέα, δεύτερον για την ύπαρξη και διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και τρίτον σε σχέση με την ικανότητα παροχής ποιότητος και καινοτομία στον τομέα αυτό. Στην αριστερά πλευρά της διαφάνειας βλέπετε στοιχεία από διάφορες πηγές για τις περικοπές που υπήρξαν. Σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα βλέπουμε περικοπή των προϋπολογισμών και από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη υπηρεσιών. Αυτό συμπεριλαμβάνει και μείωση προϋπολογισμών για άμεσες πληρωμές και για συστήματα υποστήριξης. Σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, βλέπουμε ότι στην Ευρώπη αυξάνονται οι λίστες αναμονής. Αυτό είναι αντιφατικό. Από τη μία μεριά αυξάνονται οι ανάγκες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρώπη γυράσκει, αλλά υπάρχει συγχρόνως και μείωση παροχής υπηρεσιών λόγω της περικοπής των προϋπολογισμών. Αυτό το οποίο είναι ενισχυτικό είναι ότι οι μικρές καινοτόμες υπηρεσίες πλήττονται περισσότερο από την κρίση από ότι οι πιο παραδοσιακές μορφές υπηρεσιών. Έρχομαι λοιπόν στο τρίτο στοιχείο, που είναι το στοιχείο της ποιότητας των φορέων, το οποίο έχει επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση. Σε όλη την Ευρώπη βλέπουμε την τάση να γίνεται εκ νέου ιδρυματοποίηση, η οποία φέρνει τους ε, ασθενείς και εμπλεκόμενους σε διάφορα μεγάλα κέντρα. Βλέπουμε να υπάρχει μια πορεία περιορισμού της υποστήριξης που σε άτομα ευάλωτα που είχαν δημιουργηθεί στις δεκαετίες του 40 και του 50 και επομένως απλώς δίνουν κάποια ε, τροφοδοσία σε υπηρεσίες χωρίς να δίνουν στα άτομα αυτά τη δυνατότητα να συμμετέχουν πιο πλήρως σε αυτή τη διαδικασία αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. <clears throat> Ένα δεύτερο θέμα το οποίο θα ήθελα να σας τονίσω είναι ο αντίκτυπος για αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες. Βλέπουμε ότι η οικονομική κρίση κινδυνεύει να γίνει μια πραγματική κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δυνατότητες απασχόλησης για άτομα με αναπηρίες παραγωγός χάρη είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Υπάρχει μείωση και στην ανοιχτή αγορά εργασίας και σε διάφορες περιοχές προστατευόμενης εργασίας. Δεν υπάρχουν πια προσφορές εργασίας. Τα άτομα τα οποία έχουν αναπηρίες και ήταν οι τελευταίοι που μπήκαν στην αγορά εργασίας και οι πρώτοι που εκδιώχτηκαν από αυτήν. Το θέμα της περιεκτικής παιδείας. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό εργαλείο για να έχουμε μια περιεκτική κοινωνία και να δώσουμε πρόσβαση σε μια αγορά εργασίας που είναι ανοιχτή είναι αυτό ακριβώς, η παιδεία. Υπήρξαν πολύ καλά προγράμματα σε κράτη-μέλη που προωθούσαν την ενσωμάτωση των ατόμων με μειονεκτήματα, αλλά περιεκόψαν και σταματήσαν. Το πιο λυπηρό ήταν αυτό που έγινε στην Πορτογαλία που είχε αναπτύξει ένα πολύ καλό σύστημα, το οποίο τώρα έχει διακοπεί. Η ανεξάρτητη διαβίωση, η τρίτη πτυχή της ζωής των ατόμων με αναπηρίες που είναι πάρα πολύ σημαντική. Βλέπουμε μείωση των προϋπολογισμών για άτομα με μειονεκτήματα και μέτρα να εγκλείονται σε ιδρύματα όλα αυτά τα άτομα αντί να ζουν ανεξάρτητα. Βλέπουμε λοιπόν να αναδύεται μία τάση η οποία είναι ιδιαίτερα σαφής ότι και σε αυτή την περίπτωση οι πιο καινοτόμε υπηρεσίε περικόπτονται περισσότερο από τις παραδοσιακές υπηρεσίε τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά για το κόστος που πρέπει να υπομισθούν τα άτομα με μειονεκτήματα. Καταρχήν έχουμε μη λιγότερες υπηρεσίες, είναι σαφές. Βλέπουμε επίσης όμως ότι η μερίδα του κόστους, όπως, είπε και, όπως είπαν και οι δύο προλαλήσαντες, η μερίδα του κόστους που πρέπει να επομιστεί ένα άτομο με αναπηρίες για τις υπηρεσίες αυτές έχει αυξηθεί. Είναι όλο και μεγαλύτερο αυτό το τμήμα λοιπόν του κόστους σε όλη την Ευρώπη και βλέπουμε επίσης ότι η άτυπη περίθαλψη και υποστήριξη προς τα άτομα αυτά, δηλαδή από την οικογένεια και τους κοντινούς αυτού του ατόμου, πρέπει να αναλάβει τη σκητάλη. Και εδώ τίθεται και ένα θέμα φίλου. Όταν λέμε οικογένειες, μιλάμε για τις μητέρες. Οι μητέρες κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους γιατί πρέπει να φροντίσουν τα ευάλωτα άτομα στις οικογένειές τους για τα παιδιά τους ή ακόμα και για ενήλικες που έχουν αναπηρίες. Αυτό είναι μια πολύ αρνητική, πολύ λυπηρή εξέλιξη. Και έρχομαι στην επόμενη διαφάνεια. Αυτό που βλέπουμε είναι αν θυμηθούμε την ε, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες, ξεπεράσαμε μια αρχική πατερναλιστική προσέγγιση σε μια προσέγγιση που έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρήσαμε ότι αυτοί οι οποίοι έχουν αναπηρίες έχουν κάποια ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να γίνουν σεβαστά. Ενώ η κρίση τώρα έχει αναστρέψει αυτή τη διαδικασία. Μας έχει φέρει σε μια κατάσταση που επανεχόμαστε στην αρχική πατερναλιστική προσέγγιση ότι αυτά τα άτομα δεν έχουν ικανότητες και είναι απλώς ευάλωτα και δεν πρέπει να συμμετέχουν στην αντιμετώπιση και στην κοινωνία. Είχα μιλήσει με ένα άτομο το οποίο είναι 40 λίγο χρονών και σε μια συνάντηση στην Πράγα μου είπε πριν από λίγα χρόνια με βλέπανε όλοι με ήκτο ουσιαστικά στα μάτια τους και αυτό ήταν λυπηρό. Τώρα πια μου λένε εσύ μου παίρνεις τους φόρους που πληρώνω και τις κοινωνικές παροχές και κοστίζει σε βάρος στην κοινωνία μας. Αυτή η εξέλιξη λοιπόν είναι δραματικού χαρακτήρα και δείχνει ότι αυτή η κρίση που διερχόμαστε μπορεί να έχει και μακροχρόνιο αντίκτυπο για το πώς εμείς ως κοινωνία αντιμετωπίζουμε τα άτομα με αναπηρίες και άλλα μειονεκτήματα, τα άτομα τα οποία χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη στην κοινωνία μας και περιορίζουν την δυνατότητα αυτών των ατόμων να συμμετέχουν στην κοινωνία και να απολαμβάνουν τα κοινωνικά αγαθά. Υπάρχει και αυξανόμενη ανισότητα σε ό,τι αφορά τις πρόσβα, την πρόσβαση στις υπηρεσίες. Βλέπουμε καταρχήν ανισότητα λόγω του εισοδηματικού επίπεδου, όσο πιο πολύ πρέπει να συμβάλλει κανείς σε μια υπηρεσία, παίζει και μεγαλύτερο ρόλο το εισόδημα που έχει κανείς. Επιπλέον όμως βλέπουμε αυξανόμενες ανισότητες μεταξύ διαφορών ευαλώτων ομάδων και ιδίως τα άτομα τα οποία έχουν μεγαλύτερες αναπηρίες, με πνευματικά προβλήματα, με πνευματικές αναπηρίες, βλέπουμε όλο και μεγαλύτερη ανισότητα να αναδύεται. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στις νέες ευάλωτες ομάδες που πολύ συχνά τις ξεχνάμε. Είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν τα άτομα με αναπηρίες και άλλα μειονεκτήματα ακόμα και πριν από την κρίση αυτοί οι οποίοι φροντίσανε τα άτομα με μειονεκτήματα είχαν χαμηλότερο εισόδημα από αυτούς οι οποίοι βρισκόταν σε άλλες υπηρεσίες μια διαφορά 25-30% σε, σε εισόδημα μεταξύ αυτών που βρίσκονται στον τομέα της περίθαλψης και αυτών που εργάζονται σε άλλες υπηρεσίες. Αυτό επιδεινώνεται όλο και περισσότερο. Αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στον τομέα της περίθαλψης έχουν γίνει πια οι φτω... εργαζόμενοι φτωχοί στην Ευρώπη. Και επίσης αυτοί οι οποίοι παρέχουν άτυπη υποστήριξη και περίθαλψη σε οικογενειακό επίπεδο γίνονται πιο ευάλωτοι, χάνουν τη θέση τους εργασίας, μπορεί να χάσουν το εισόδημά τους, μπορεί να καταλήξουν να μπουν στο χώρο της ένδυας. Η κοινωνική καινοτομία τώρα. Στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Ολλανδία, στην Ουγγαρία, Γαλλία, Γερμανία υπήρξαν νέες, ε, νέα υποδείγματα καινοτόμων υπηρεσιών περίθαλψης από δημόσιους φορείς, από ΜΚΟ κτλ. Οι περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες σταμάτησαν να εξελίσσονται λόγω της κρίσης. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση ήταν ένα πραγματικό πρόβλημα για όλους αυτούς τους φορείς. <clears throat> Και τώρα ζητάμε να υπάρξει καινοτομία Μα πρέπει να πω ότι στο δικό μου τομέα υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την συνθηματολογία που έχει να κάνει με την καινοτομία. Γιατί είναι σύνθημα μονάχα αλλά χωρίς πολύ περιεχόμενο. Έχουμε την εντύπωση στο δικό μου τομέα ότι πρώτα σφάζουμε το κοτόπουλο και τώρα ζητάμε Προσφάσουμε πρώτα την κότα και μετά ζητάμε να κάνει περισσότερα αυγά και καλύτερα αυγά. Υπήρχε καινοτομία στον τομέα αυτό. Τα μέτρα λιτότητα όμως σε κάποιε από τι χώρε ή στι στις περισσότερες τη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής έχουν <coughs> ανακόψει αυτή τη θετική εξέλιξη. Για μας είναι σημαντική λοιπόν η κοινωνική καινοτομία και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την πρωτοβουλία τη Κομισιόν και του, και του Κοινοβουλίου στα θέματα αυτά. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με περικοπές χρηματοδότηση. Θα πρέπει να σκεφτούμε την ποιότητα των υπηρεσιών, την περιεκτικότητά τους, τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ατόμων με μειονεκτήματα και των άλλων ευάλωτων ομάδων. Τελευταία μου ε, διαφάνεια, ελπίζω να έχω κάποια δευτερόλεπτα, έτσι θα είναι κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν διάφορες επιλογές εδώ. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είναι κεφαλαιόδες η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι φορείς της να σταθμίσουν μια σαφή θέση σε σχέση με τα αποτελέσματα της κρίσης για τον τομέα περιθάλψης και τον αντίκτυπο των περικοπών στη χρηματοδότηση περιθάλψης. Και η Κομισιόν, μπορεί να το κάνει και η Επιτροπή σας και το Σύνολο Κοινοβούλιο. Καταρχήν μπορούμε, μπορείτε να υποστηρίξετε το ψήφισμα αυτό το οποίο υποστηρίζεται. Επίσης μπορεί το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει υπηρεσίες οι οποίες έχουν ευφύ χαρακτήρα και να μην ε, υποστηρίξει δραστηριότητες που περικόπτουν την ενεργή συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Το κοινωνικό πακέτο για συμπερίληψη θα πρέπει να αντιμετωπίσει την διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα των υπηρεσιών και των συστημάτων υποστήριξης. Θα πρέπει να υποστηρίξει την καινοτομία στο επίπεδο βάσης, κυρίως στο επίπεδο βάσης. Γιατί αυτό που κάνει μια υγειονομική υπηρεσία διαφορετική από μια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ότι είναι βαθιές οι ρίζες της της ε, περίθαλψης στην κοινωνία και είναι απαραίτητο για να υπάρξει ένα πραγματικό σύστημα υποστήριξης. Μια πέμπτη μορφή προσέγγισης και υποστήριξης θα πρέπει οι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απελευθερώσουν τη δυνατότητα του τομέα παρέχει θέσεις απασχόλησης. Αυτή τη στιγμή θα μπορούμε να βρούμε νέους οι οποίοι θέλουν να εργαστούν στον τομέα αυτό γιατί είναι αρνητικές οι συνδίκε εργασία Είναι σημαντική η ελκυστικότητα του τομέα και ο κοινωνικό διάλογο για τα θέματα αυτά. Ξέρει το Κοινοβούλιο ότι υπάρχει μια Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου για του κομμωτέ και τι κομμότριε, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχο αντίστοιχη επιτροπή για το κοινωνικό τομέα όπου υπάρχουν χιλιάδες περισσότεροι εργαζόμενοι. Υπάρχει ένα πρόβλημα και οι ευρωπαϊκοί φορείς θα πρέπει να βοηθήσουν να υπάρξει κοινωνικός διάλογο και σε αυτό το τομέα. Τέλος, να χρησιμοποιηθεί και ο ερευνητικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καινοτομία που βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία και ελπίζω ότι αυτά που σας είπα σας έχουν βοηθήσει στη συζήτησή σας και ελπίζω ότι θα μπορέσει το Κοινοβούλιο να είναι ένας σύμμαχός μας για να αντιμετωπίσουμε τα αποτελέσματα της κρίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ανακεφαλαίωση που κάνατε. Βλέπετε ότι σε αυτή την Επιτροπή το θέμα αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως και θα φροντίσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα αυτό. Επόμενος ε, προσκεκλημένος, ο κύριος Goodwin, ε, γραμματέας της Eurocares. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία. Πρώτα απ' όλα, να συμφωνήσω με όσους πήραν το λόγο προηγουμένως στο πάνελ. Θα συμφωνήσω λίγο πολύ με όλα όσα είπαν και δεν θα τα επαναλάβω. Εγώ εκπροσωπώ τους ανεπίσημους ε, φροντιστές, φροντίζοντες της οικογένειας, τα μέλη της οικογένειας που φροντίζουν ανθρώπους που πάσχουν από χρόνιες νόσους και παραμένουν στο σπίτι σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι αυτό το είδος φροντίδας εκπροσωπεί το 80% της φροντίδας συνολικά στην Ευρώπη. Είτε μιλάμε για θεσμική είτε νοσοκομιακή. Η συντριπτική πλειονότητα φροντίδας παρέχεται από μέλη της οικογένειας στον, στο σπίτι. Στην Ιρλανδία εκτιμούμε σε 4 δις ευρώ ετησίως ε, την αξία της φροντίδας αυτής, ενώ σε 120 δις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μιλάμε για μεγάλο ε, μερίδιο. Οι κοινωνικές, ε, τα κοινωνικά συστήματα θα μπορούσαν να καταρρεύσουν εάν αυτοί οι άνθρωποι που φροντίζουν τους αρρώστους δεν παρήχαν τις υπηρεσίες τους. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους αυτούς ουσιαστικά μπορεί να είναι αμοιβόμενοι. Εφόσον λοιπόν τους χάσουν οι εργοδότες τους, ε, είναι με καταστροφικές οι συνέπειες τα, οι εξελίξει στην οικονομία επηρεάζει τόσο αυτού που παρέχουν τη βοήθεια, όσο και αυτού που του απασχολούν, όσο και τα άτομα τα οποία χρήζουν βοήθεια. Θα υπάρξει θεσμικό πρόβλημα εάν αυτοί που φροντίζουν τα άτομα με χρόνιε παθήσει δεν μπορούν να παράσχουν την φροντίδα αυτή. Και πολλές φορές υπάρχει αντίφαση μεταξύ της ανεπίσημης φροντίδας που παρέχουν και της αμοιβόμενης εργασίας τους. Επίσης κάποιες φορές πρέπει να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις και μεταξύ διαφορετικών συνόρων. Εάν το δούμε λοιπόν από την άποψη εργαζομένου εργοδότη, οι φροντίζοντες αυτοί θα πρέπει να τύχουν κάποιας ε, μέρημνας. Παρέχουν φροντίδα υψηλού επίπεδου 80 και περισσότερες ώρες την εβδομάδα, αλλά και κάποιοι άλλοι 24 ώρες το 24ωρο, διότι το άτομο το οποίο φροντίζουν έχουν, πρόβλημα, έχουν προβλήματα συμπεριφοράς ή δυσκολίες στον ύπνο. Και αυτό αφορά ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που παρέχουν φροντίδα. Είναι λοιπόν ε, περίπλοκο το θέμα της ε, φροντίδας. Προηγουμένως αναφέρθηκε η διάσταση των φύλων. Το επίπεδο της φροντίδας ως προς την χρονική διάσταση και ως προς το περίπλοκο χαρακτήρα αφορά κυρίως γυναίκες που παρέχουν φροντίδα. Είναι σημαντικό το στοιχείο αυτό. Μιλάμε για γυναίκες που χάνουν την επίσημη εργασία τους διότι πρέπει να μείνουν στο σπίτι για να δώσουν ε, φροντίδα υψηλού επίπεδου, να στηρίξουν αρρώστους και βεβαίως έτσι αυξάνονται και τα ποσοστά φτώχειας. Η μετάβαση από τη θεσμική φροντίδα στην νοσοκομιακή και στην οικιακή φροντίδα είναι κάτι που ουσιαστικά δυσκολεύει τους ε, ανθρώπους που φροντίζουν αρρώστους. Για τα νοσοκομεία εκτάκτων περιστατικών, οι διαδικασίες τους ε, διαρκώς βελτιώνονται. Όσοι εισάγονται, παραμένουν για λίγο, κάνουν κάποια τεστ, κάποια σύντομη περίθαλψη, κάποια εγχείρηση, αλλά τείνουν να παραμένουν ελάχιστο χρονικό διάστημα ε, στα νοσοκομεία για βαριά περιστατικά. Τα τεστ γίνονται πολλές φορές την πρώτη μέρα εισαγωγής. Αυτό σημαίνει ότι την υπόλοιπη περίθαλψη την αναλαμβάνει ο άνθρωπος που φροντίζει ανεπισήμως τον άρρωστο. Ακόμα και η περίοδος παραμονής στην αντατική να συντομεύεται. Οπότε, αυτό απαιτεί ε, πόρους. Έπειτα τα νοσοκομεία βαρέων περιστατικών πρέπει να ελευθερώνουν πιο εύκολα κλίνε ώστε να παρέχουν και περισσότερες υπηρεσίε στους καταναλωτές. Την προτεραιότητα την δίνουν ε, σε αρρώστους εφόσον ελευθερωθούν κλίνε σε κάποια νοσοκομεία. Αλλά αυτό δεν είναι αναλογικό με τις ανάγκες. Άρα ο υπεύθυνο ή ο συγγενής θα πρέπει να παράσχει ακόμη φροντίδα. Έρχεται μετά το νοσοκομείο των βαρέων περιστατικών. Εφόσον το νοσοκομείο κρίνει ότι ο συγγενής δεν μπορεί να εισαχθεί. Αυτό είναι και μια μορφή εκμετάλλευση των ανθρώπων που φροντίζουν ανεπισήμω του αρρώστου. Αλλά να δούμε τι γίνεται και με τα γυροκομεία, τα οποία του οίκου ευγυρία που και αυτά τείνουν να παράσχουν υψηλού επίπεδου υγειονομική περίθαλψη. Και αυτοί ελευθερώνουν κλίνε για άλλου είδου φροντίδα ε, που κάποιε φορέ μπορεί να είναι συμπληρωματική τη φροντίδα που παρέχεται στο σπίτι. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι οι οίκοι ευγυρία ε, πιέζονται για να δίνουν υψηλότερο επίπεδο υπηρεσίε με χαμηλότερο προπολογισμό. Και αυτό δημιουργεί δυσκολίε. Οι άνθρωποι που φροντίζουν επισήμω του αρρώστου τείνουν να μην δουλεύουν σε οίκους ευγυρία ακριβώς γιατί θα χρειαζόταν ειδική μέρημνα. Κάποιοι άρρωστοι τις φροντίδα που χρειάζονται την λαμβάνουν, τη φροντίδα που χρειάζονται τη λαμβάνουν και στο σπίτι. Έτσι, η φροντίδα τίνει να παραμείνει ανεπισήμως στο σπίτι παρά να περάσει σε αμοιβόμενο πλαίσιο, στους οίκους ευγυρίας, λόγω χάρη. Κάτι άλλο που αλλάζει και το καλωσορίζουμε θερμά είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις. Επιτρέπει στους ανθρώπους να παραμείνουν στο σπίτι τους, να μειώσουν τις επισκέψεις τους στο νοσοκομείο και να πάνε στα τοπικά κέντρα υγείας χάρη στις τεχνολογικές αλλαγές. Αυτό βελτιώνει την κατάσταση και του ασθενούς και του ίδιου του υπευθύνου της φροντίδας. Υπάρχουν υπηρεσίες υποστήριξης λοιπόν χάρη στα τεχνολογικά μέσα. Βεβαίως ε, οι παράγοντες που τα επηρεάζουν όλα αυτά είναι οικονομικοί. Και οι ανεπίσημοι φροντι... φροντίζοντες τους αρρώστους είναι σαν να είναι μια αυτόματη επιλογή. Γι' αυτό έχει αυξηθεί το επίπεδο φροντίδας στο σπίτι. Αυτή ήταν μια σημαντική παρατήρηση. Η επόμενη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι το επίπεδο φροντίδας. Το επίπεδο φροντίδας γίνεται όλο ένα και πιο περίπλοκο στο σπίτι. Πρώτα απ' όλα τα φάρμακα. Κάποιε φορέ οι ασθενεί που επιστρέφουν στο σπίτι του μετά από νοσοκομιακή περίθαλψη έχουν ιδιαίτερα περιπλοκή συνταγογράφηση και με χρήση τεχνολογικών μέσων και με διαδικασίε πολύ περίπλοκε, όπω η αιμοκάθαρση λόγου χάρη. Και με ελάχιστη στήριξη. Όταν εδώ δημιουργούνται προβλήματα, θα πρέπει την λύση να τη βρουν μόνοι τους αυτοί οι άνθρωποι που φαντίζουν επισήμως τους συγγενείς. Είδαμε πρόσφατα ένα, ένα περιστατικό όπου ο άνθρωπος που ε, παρήχε τη φροντίδα σε ηλικιωμένη κυρία ήταν ένα συγγενής με ειδικέ ανάγκες και κάποια στιγμή έπρεπε να εισαχθεί και ο ίδιος στο νοσοκομείο. Δεν μπορούσε κανείς να διευκολύνει ε, την ε, κατάσταση αυτή. Έπρεπε η ίδια να εξεύρει τα μέσα, να απευθυνθεί σε φίλους, σε συγγενείς, ε, στην κοινωνική πρόνοια για να στηρίξουν την άρρωστη που θα έμενε μόνη. Ήδη όμως εκείνη παρέχει πλήρη φροντίδα στο σπίτι σε μια ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ η ίδια υποφέρει από βαριά αναπηρία. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι σε αυτό το το οποίο πριν υπάρξουν οι γνωστές περικοπές είχαμε ήδη την κατάσταση που περιέγραψα και που τώρα έχει επιβαρυνθεί πολύ. Υπάρχουν περικοπές εφόσον η κυβέρνηση λόγου χάρη αποφασίζει ότι θα μειώσει τους πόρους προς τους ε, φροντιστές. Κάποτε γινόταν μια αξιολόγηση βάσει των ωρών φροντίδας που πρόσφεραν στο σπίτι. Αυτή τη στιγμή όμως η φροντίδα αποτιμάται με τρόπο πολύ επιφανειακό. Μπορεί οι ώρες να έχουν αυξηθεί μέσα σε μια τριετία, αλλά θα προσπαθήσουν οι αρχές να δώσουν στήριξη σε κάποιον που μπορεί να μην παράσχει πάρα πολύ λίγη φροντίδα και έτσι μοιράζεται λιγότερο δίκαια το κονδύλι και ασκείται μεγαλύτερη πίεση στου ανθρώπους αυτούς που υποστηρίζουν τους αρρώστου. Υποφέρουν πολλές φορές από άγχο ή και κλινική κατάθλιψη οι άνθρωποι αυτοί λόγω της πίεσης που τους ασκείται. Επίσης υπάρχει μείωση των δωρεών που γίνονται στου ανθρώπους αυτούς των επιδομάτων και των κονδυλίων που προβλέπονται για βασικές αλλαγές, προσαρμογές του χώρου του σπιτιού για να μπορέσει να προσαρμοστεί στι ανάγκε των αρρώστων. Λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να γίνουν δικαιούχοι ιατρικών καρτών δελτίων και η περίοδος αξιολόγησης και εξέτασης της αίτησής τους κρατάει πολύ περισσότερο πλέον. Επιπλέον, όσοι έχουν δικαίωμα επιστροφής κάποιων εξόδων φαρμάκων, Κάποιες φορές έχουν ε, τριπλασιάσει την εισφορά τους σε σχέση με το κόστος που τους καλύπτουν. Επίσης να μιλήσω για τα σωρευτικά φαινόμενα. Διότι σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο δεν υπάρχει καλή συνεργασία. Κάποιοι εισάγονται σε νοσοκομείο λόγω ενός, βαριού, ενός έκτακτου περιστατικού όπως ένα κεφαλικό αλλά γρήγορα επιστρέφουν σπίτι πλέον, όπου το μέλος της οικογένειας θα πρέπει να αποκτήσει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να φροντίσει τον άρρωστο, με πολύ μεγάλες απαιτήσει. Οι προσαρμογές επίσης πρέπει να γίνουν στο χώρο του σπιτιού, δεν μπορούν να καλυφθούν από τα επιδόματα που δίνονται. Οπότε πολλές φορές λένε στους ανθρώπους αυτούς είσαστε στον κατάλογο για να λάβετε βοήθεια για του χρόνου. Αλλά είναι πολύ αργά μέχρι την επόμενη χρονιά και αυτό είναι απέσιο εάν σκεφτεί κανείς ότι αυτό συμβαίνει σε μια κοινωνία όπου οι επίσημοι φορείς έχουν προβλεπόμενους πόρους, οι υπάλληλοι έχουν τους μισθούς τους, αλλά δυστυχώς δεν κατευθύνουν τις βοήθειες εκεί που είναι πλέον απαραίτητες. Την πίεση ουσιαστικά την ταβάνε οι ίδιοι άνθρωποι που φροντίζουν τους αρρώστους. Κάποιες φορές μάλιστα οι υπηρεσίες και τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών καθυστερούν υπέρμετρα. Και αυτό έχει γίνει και όπλο στρατηγικό για να γίνονται από εξοικονομήσεις χρημάτων. Γίνονται διαρκώς αιτήσει επί αιτήσεων λοιπόν από τους ανθρώπους αυτούς για να λάβουν τα χρήματά τους, αλλά καμιά φορά καθυστερούν 6 μήνες μέχρι και 2 χρόνια. Πρόεδρος, με συγχωρείτε αν μπορείτε να ολοκληρώσετε για να έχουμε και ερωτήσεις. Ναι, βλέπουμε περιπτώσεις όπου κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν ακόμη να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για αρρώστους με ακράτεια και πρέπει να απευθυνθούν ε, στην καλή θέληση κάποιων νοσοκόμων από νοσοκομεία. Πραγματικά σας παρακαλώ συντομεύσετε, διότι έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Εάν μπορείτε, συντομεύστε. Δύο-τρεις σύντομες παρατηρήσεις μόνο. Πρώτον, νομίζω ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη στοιχείων. Οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε για να διευκολύνετε την μελέτη των θεμάτων αυτών και να έχουμε δεδομένα θα ήταν καλό. Η Eurostat μπορεί να διαγραμματίσει εδώ σημαντικό ρόλο, διότι σε κάποιες χώρες έπρεπε να ζητηθούν συγκεκριμένα στοιχεία για το ρόλο των ανεπίσημων αυτών ανθρώπων που φροντίζουν τους αρρώστους, των ανεπίσημων βοηθών των αρρώστων και να εντοπιστούν συγκεκριμένε καταστάσει, να αποφύγουμε τι ορευτικέ συνέπειε δηλαδή σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Αυτό θα ήταν μια σημαντική συμβολή. Και αυτό που θα είχα να σα πω είναι ότι ό,τι μπορείτε να κάνετε για να αναπτυχθεί μια συνολική πολιτική δράση ώστε τα κράτη να ενθαρρυνθούν να δημιουργήσουν στρατηγικές για τους ε, ανθρώπου που φροντίζουν τους αρρώστους ήδη θα ήταν αρκετό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Θα δώσω το λόγο στον Αλεχάνδρο Σέρκας που ζήτησε το λόγο. Και μετά... ποιο άλλο, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας πω καταρχήν ότι σας άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία και μεγάλη συγκίνηση συγχρόνως γιατί ο μόνος τρόπος να έχουμε πραγματικά επιχειρήματα και να έχουμε συγκεκριμένα πρόσωπα αυτή τη στιγμή έναντι αυτού του εφιάλτη που ζούμε στην Ευρώπη, πως καταστρέφεται η συμβίωση των ανθρώπων στην Ευρώπη, είναι να έχει τα στοιχεία σε αυτά. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο και να σας θέσω και κάποια ερωτήματα. Εγώ έρχομαι από την Ισπανία. Η Ισπανία ήταν ένα εργαστήριο κατά κάποιο τρόπο όπου μπορεί να δει κανείς όχι τα αποτελέσματα μόνο της κρίσης αλλά και του τρόπου με τον οποίο έγινε η διαχείριση της κρίσης. Υπήρξαν πολιτικές αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν που είχαν αποτελέσματα για τους απλούς ανθρώπους. Θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικές αυτές οι αποφάσεις, να μην είναι αυθαίρετες παραγωγός χάρη, το να χαθεί η δυνατότητα μεταφοράς των ε, αρρώστων που πηγαίνουν για αιμοδιάλυση. Αυτό σίγουρα δεν βοηθάει όλα αυτά τις χιλιάδες ατόμων που βρισκόνται σε αυτήν την κατάσταση. Η κρίση λοιπόν ήταν απλώς ένα άλοθη για να εφαρμοστούν αποφάσεις όπως αυτή της ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά των δημοσίων υπηρεσιών και ιδιαίτερα της περίθαλψης. Βλέπουμε στην Ισπανία λοιπόν όχι μόνο μία τελείως ανίκανη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Βλέπουμε την κατάλυση της αρχιτεκτονικής και των αξιών του συστήματός μας. Το σύστημα στην Ισπανία βασιζόταν στο δικαίωμα κάθε πολίτη να την χάνει περίθαλψη. Τώρα πια μόνο αυτοί που είναι ασφαλισμένοι και έχουν λεφτά στην τσέπη τους μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες ακόμα και αν ζητάει κανείς ένα ευρώ για συμβολή του ασθενού, αυτό είναι παράλογο για κάθε ασθενή που δεν έχει λεφτά καθόλου, που είναι άνεργο. Δεν μπορεί να πληρώνει για κάθε φάρμακο που παίρνει ένα ευρώ. Αυτές είναι πολιτικές επιλογέ λοιπόν που στοχεύουν στο να καταστρέψουν την αρχιτεκτονική ενό συστήματο που βασίζεται στα δικαιώματα των ανθρώπων. Και μια κίνηση προς την εμπορευματοποίηση της υγείας και των φαρμάκων. Αν λοιπόν κάποτε περάσει η κρίση και συνεχίσει αυτή η προσέγγιση, θα έχουμε και πάλι, θα έχουμε στις, και πάλι το πρόβλημα αυτό στη συνέχεια. Γιατί καταστρέφηκαν δομέ. Υπήρξε μια διαρθρωτική αντιμετώπιση ιδεολογικού χαρακτήρα για να καταληθεί το σύστημα. Το ερώτημά μου είναι ποιο θα είναι το κόστος που θα προκύψει για τη δημόσια υγεία. Όλη αυτή η καταστροφή δεν θα είναι δωρεάν. Όταν χιλιάδες και εκατομμύρια ανθρώπων πάψουν να έχουν δωρεάν περίθαλψη. Βλέπετε να αναδύονται νέα προβλήματα, προβλήματα φυματίωσης παραδείγματο χάρη ή άλλων ε, χρονίων ασθενειών που δεν αντιμετωπίζονται αυτή τη στιγμή και μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα ε, μεταδοτικών ασθενειών και άλλων προβλημάτων. Τι κόστος θα έχει τελικά αυτή η διαδικασία εξοικονόμησης μέσα εισαγωγικά και για τις δημόσιε υπηρεσίες υγείας και για μας. Και βλέπετε τι γίνεται στην Ελλάδα στην Πορτογαλία, σε άλλες χώρες πώς καταστρέφεται η υγειονομική περίθαλψη. Υπάρχουν επίτροποι οι οποίοι επικροτούν τα μέτρα αυτά. Λοιπόν, πώς το βλέπετε εσείς αυτό. Ήδη στην Ισπανία έχει υπάρξει μια αναδυόμενη συνένεση από όλου του εργαζόμενου στο υγειονομικό τομέα ότι αυτό δεν είναι μια κομματική τοποθέτηση, μια πολιτική επιλογή. Είναι μια πορεία καταστροφή τη ίδια τη Ευρώπη. Πώ λοιπόν μπορεί να φτάσει η φωνή αυτή ε, των οργανώσεών σα στου φορεί τη Ευρώπη. Μέρφυ και η κυρία Άρκιν μετά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, τέσσερις ομιλητές, ε, διότι νομίζω διέδωσαν μια πάρα πολύ καλή εικόνα των επιπτώσεων της πολιτικής λιτότητας στην Ευρώπη, ε, σε βασικά δικαιώματα, σε υγειονομική περίθαλψη, πώς αφαιρούνται δικαιώματα. Και είδαμε πώς επηρεάζονται συγκεκριμένες ομάδες, οι αποκαλούμενες ευάλωτες ομάδες. Αλλά δεν είναι ευάλωτες επειδή οι ε, υποφέρουν από κάτι των γενές, απλά επειδή η κοινωνία τους ε, αντιμετωπίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εκείνο που με εντυπωσίασε είναι ότι αναφέρατε πολλές και σημαντικές επιθέσεις στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αναφερθήκατε σε περικοπές, σε άμεσες, άμεσα επιδοτήματα, ενίσχυση στη θέση εργασίας και πολλά άλλα. Και κάθε ένα από αυτά είναι πολύ σημαντικά. Όμως το σημαντικότερο είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για σόρευση περικοπών, αλλά πρόκειται και για την διαφορά στην ποιότητα ζωής μοιάζει δηλαδή να υπάρχει σημαντική επιδείνωση της ποιότητας της ζωής ε, των ατόμων με αναπηρία. Είχαμε προχωρήσει κάπως και τώρα ε, οπισθοχωρούμε σε, ένα, σε μια άλλη μορφή και σε όλα αυτά τα προβλήματα της ε, ιδρυματοποίησης. Εδώ πρέπει να αντισταθούμε. Και δεύτερη παρατήρηση. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι αυτά τα άτομα είναι θύματα αλλά επίσης πρέπει να γνωρίσουμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος, δηλαδή σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη αυτές ε, οι ευάλωτες ε, ομάδες αγωνίστηκαν ε, κατά της ε, πολιτικής λιτότητας στην Ιρλανδία. Αυτή είναι η πρώτη που κινητοποιήθηκαν κατά κάποιων ε, περικοπών και μετά βοήθησαν στο να προκύψουν μεγαλύτερα κινήματα κατά της λιτότητας. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποδώσει δικαιοσύνη ή η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζονται οι ευάλωτοι είναι να ε, συγκεντρωθούν με άλλους ε, στην Ευρώπη και επίσης ε, τα θέματα αυτά να εξεταστούν στο σύνολό τους από τα συνδικάτα, να καταστούν δηλαδή τμήμα του μεγαλύτερου αυτού αγώνα. Η αντίδραση είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντισταθούμε στην περικοπή δικαιωμάτων και να διεκδικήσουμε περισσότερα. Η κυρία Χάρκιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο Κοινοβούλιο πάντοτε ευχαριστούμε τους ε, προκεκλημένους μας για τις εισηγήσεις τους. Αλλά εσάς σας ευχαριστώ από καρδιάς, διότι πραγματικά με εντυπωσίασαν όσα μας είπατε και εντυπωσιάστηκα περισσότερο από ό,τι συνήθω. Διότι το θέμα δεν είναι να μιλήσετε απλώ για την κατάσταση. Εσεί μα κάνατε και κάποιε προτάσει. Και αυτό ακριβώ για μα είναι πολύτιμο ε, για το ρόλο μα ω ε, βουλευτών. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν. Εάν είναι διαθέσιμε οι παρουσιάσει σα, εγώ πραγματικά θα τις ήθελα. Κράτησα κάποιε σημειώσει, δεν τα έγραψα όμω όλα να συμφωνήσω με τον συνάδελφο Πολ Μέρφυ εν μέρη, όχι πλήρως. Εκείνος δεν πιστεύει ότι θα σας δικαιώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που κι εμείς μπορούμε να κάνουμε και εσείς μας δώσατε κάποιες ιδέες. Μιλήσατε για πράγματα όπως ο επίπεδο των μισθών ή ο κοινωνικός διάλογος. Αυτό είναι ένας χώρος όπου μπορούμε να διαδραματίσουμε κάποιο ρόλο, να έχουμε κάποια επιρροή και Ειδικά σήμερα με το νέο μας ρόλο έχουμε αμεσότερη επιρροή. Μια δυο ερωτήσει και θα είμαι πολύ σύντομη στα σχόλιά μου, Πρόεδρε. Είπατε για τα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα. Διάβασα κάποια δημοσιεύματα γι' αυτό και η ερώτησή μου είναι πώς τα πάει ο κόσμος, πώς επιβιώνει τα καταφέρνουν. Για τον κύριο από τη Γαλλία, μιλήσατε για οικουμενική γεωνομική περίθαλψη και την ασφάλιση που έχει προβλεφθεί. Έχει βοηθήσει καθόλου το σύστημα αυτό, έχει κάνει κάποια διαφορά. Και για τον κύριο από το Βέλγιο, νομίζω ότι ήταν πραγματικά η παρέμβασή σας δραματική, ιδίω στην παρατήρηση για το πώ αντιλαμβάνονται σήμερα οι υπόλοιποι πολίτε, του ανθρώπου με του ειδικέ ανάγκε. Χρειάστηκε πάρα πολλή χρόνο για να αλλάξουν αυτέ οι προκατάληψει και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από τη μια μέρα στην άλλη, σχεδόν βλέπουμε του ανθρώπου με ειδικέ ανάγκε. Όπω εσεί μα είπατε, υπάρχει μια τάση να συμβαίνει αυτό πάντω. Έχετε ενδείξει. Μάλλον νομίζω ότι υπάρχουν ενδείξει ότι πρέπει να αναλυθεί άμεση δράση για το θέμα αυτό, περισσότερο από ότι για άλλα. Ίσως η κοινωνική καινοτομία, η ιδέα του κοινωνικού διαλόγου σε συγκεκριμένου τομεί να είναι ε, μια ιδέα. Και για τον κύριο Γκούντουιν από του γύρω κέρες, μιλήσατε για τα μέλη τη οικογένεια που φροντίζουν αρρώστου. Κάποιε φορέ αναλαμβάνουν και ιατρικά καθήκοντα οι άνθρωποι αυτοί. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να προτείνουμε στα κράτη-μέλη τι στρατηγικές να διαμορφώσουν για αυτούς τους ανθρώπους, για όσους φροντίζουν αρρώστους στα σπίτια τους. Σας ευχαριστώ και πάλι, και πάλι ιδιαίτερος για τις συζητήσει σας. Ε, Κυρία Λάμπερτ, θέλετε να σχολιάσετε. Με συγχωρείτε. Έτσι κι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε στα αγγλικά. Λέει η πρόεδρος. Έχουμε 10 λεπτά με ένα τέταρτο. Θα ζητήσω όμως από τον κύριο Λεγκρό εφόσον γνωρίζει τι έγινε στη Γαλλία, να μας πει τι πιστεύει ότι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μα είπατε πολλοί από εσά το, το ότι υπάρχει πρόβλημα με τα δεδομένα. Είναι μια σοβαρότατη πτυχή αυτή. Την έχουμε εντοπίσει. Στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020 έχουμε όμως υπόψη το θέμα αυτό. Για τα ζητήματα καταπολέμησης της φτώχειας δεν έχουμε ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων. Κύριε Λάμπερτ. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ με αυτούς ε, που είπαν σήμερα ότι πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Αυτά που λέτε είναι συγκεκριμένα, να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά ίσως θα πρέπει να βρούμε και κάτι για το μέλλον. Ένα λοιπόν από τα θέματα που με απασχολημένα είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για ε, τα φάρμακα, το κόστος δηλαδή της ε, του ασθενούς. Ακόμα και το ίδιο το κόστος των φαρμάκων. Το κόστος είναι πολύ ψηλό. Είναι πολύ ακριβά τα φάρμακα δεν ξέρω αν αυτό είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής μας, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ε, γίνονται οι διαγωνισμοί φαρμάκων. Και όσον αφορά τον εθελοντισμό, θέλω να πω ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο οι εθελοντές να επικρίνουν αυτά τα οποία διαδραματίζονται γιατί εμπλέκονται και αυτή, σε αυτή την ε, όλη κατάσταση όσο εξελίσσεται. Θα ήθελα να έχω λοιπόν τα σχόλιά σας επ' αυτού. Ε, Ευχαριστούμε. Να δώσουμε και πάλι το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Με τη σειρά με την οποία πήραν το λόγο, ο κύριος Κανάκης πρώτα. Εάν μπορείτε, τρία-τέσσερα λεπτά η απάντησή σας. Προσπαθήσω να είμαι απολύτως συγκεκριμένος. Ε, καταρχήν σε σχέση με το, με την, το ερώτημα για τις νέες ασθένειες που βλέπουμε. Ξαναβλέπουμε στην Ευρώπη ασθένειες που τις είχαμε ξεχάσει. Πιστεύαμε ότι δεν θα επέστρεφαν. Για παράδειγμα, η φυματίωση. Ξαναβλέπουμε σύφυλλη. Ειδικά για τη φυματίωση υπάρχει ένα θέμα, μια και είναι η νόσος των φτωχών. Ότι πολλές φορές, ε, περιπτώσεις όπως στην Ελλάδα, κρύβουμε το πρόβλημα ή αγνοούμε ότι το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα δημόσια υγεία. Στην Ελλάδα στοχοποιήσαμε όπω και στο AIDS του ανθρώπου που ήταν φορεί. Έγινε το πρωτοφανέ στην Ελλάδα να δείξουμε στην τηλεόραση τα θύματα με AIDS που κατηγορούνταν για πορνεία κατηγορώντα ουσιαστικά τα θύματα και γυρίζοντα την ιατρική ηθική πολύ πίσω. Ξεχνάμε ότι αν κάποιο έχει φυματίωση, για παράδειγμα, μπορεί να κολλήσει κάποιο άλλο πάρα πάρα πολύ εύκολα σε ένα μέσο δημόσια υγεία. Η δημόσια υγεία δεν σχετίζεται με τα διοικητικά δικαιώματα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Θα έλεγα ότι μια πολύ μεγάλη συνέπεια που θα έχουμε θα είναι μια μείωση του προσβόκιμου επιβίωση στι χώρε του Νότου. Στην Ελλάδα το περιμένουμε. Φοβάμαι ότι δεν θα μπορούμε να το ιδεολογήσουμε γιατί ότι οφείλεται στα μέτρα λιτότητα που είναι, διότι άνθρωποι που δεν παίρνουν πια τα φάρμακά του ή δεν έχουν πρόσβαση σε μια κανονική διατροφή, δεν μπορεί κανένα να τα αποδείξει, αλλά είναι κάτι, θα έλεγα, που το περιμένουμε. Έχουμε ένα παράδειγμα σε σχέση με του εμβολιασμού αναφορικά με τα κρούσματα μίσλ, τα οποία είχαμε στην Ευρώπη 30.000, η έρευνα των γιατρών του κόσμου σε όλη την Ευρώπη έδειξε ότι 8 στους 10 που είχαν προσληφθεί ήταν ανεμβολίαστοι. Άρα λοιπόν αν υπήρχε ένα πρόγραμμα καθολικού εμβολιασμού και ο εμβολιασμός πρέπει να αφορά τους πάντες, χωρίς διακρίσεις, γιατί είναι ένα θέμα υγείας θα είχαμε αποφύγει αυτά τα κρούσματα ε, στην Ευρώπη και κατά συνέπεια και το κόστος τέλος σε σχέση με το πώς περνάει ο κόσμος στην Ελλάδα και ποια είναι η κατάσταση. Πρέπει να σας πω πάρα πολύ δύσκολα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δημιουργώνεται στους πιο φτωχούς ανθρώπους ένας τέταρτος κόσμος. Ένας τέταρτος κόσμος φτώχειας ανθρώπων οι οποίοι δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Σας λέω μόνο ότι κάθε μέρα η ηλεκτρική εταιρεία κόβει χίλιες συνδέσεις ρεύματος. Έχουμε βρεθεί σε σπίτια ηλικιωμένων οι οποίοι δεν έχουν ρεύμα πια, δεν έχουν νερό, πηγαίνουν στα συσίδια για να βρουν τρόφιμα, ουσιαστικά εκλυπαρούν για λίγα φάρμακα. Το χειρότερο από όλα δεν είναι η εικόνα αυτή. Το χειρότερο είναι ότι αυτό τίνει να γίνει μόνιμο, δημιουργώντα τον κόσμο την αίσθηση μια αδικία μόνιμη, η οποία βέβαια θα οδηγήσει σε πολιτικέ συμπεριφορέ αντίστοιχε, οι οποίε θα είναι τελείω αντιευρωπαϊκέ. Εκείνο λοιπόν που ζητάμε από εσά δεν είναι μόνο μια παρέμβασή σα και μια πίεσή σα για να γίνει κατανοητό ότι τα μέτρα λιτότητα που πιθανόν πρέπει να υπάρχουν σε χώρε που έχουν προβλήματα όπω η Ελλάδα δεν θα πρέπει να στοχεύουν μόνο του πιο φτωχού και αυτού που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το δημόσιο σύστημα υγεία. Αλλά θέλουμε και τη βοήθειά σας, διότι ο λόγος σας μετράει στις χώρες και στους πολίτες και στις κυβερνήσεις των χωρών να γίνει αντιληφτό ότι δεν μπορούμε να χτίζουμε μια κοινή Ευρώπη αλληλεγγύης όταν τους πιο φτωχούς, τους ταπεινούς και τους καταφρονεμένους συστηματικά τους αποκλείουμε. Πρέπει να ξαναμπεί στην ατζέντα το θέμα των δικαιωμάτων των πιο φτωχών ανθρώπων και η υγεία είναι το πιο χαρακτηριστικό πεδίο αυτών των δικαιωμάτων. Ε, Ωραία. Τέσσερα σημεία για να συμπληρώσω αυτά που ελέγχθησαν. Είμαι μέσα στους, ε, στο δίκτυο των εμπειρογνώμων που εργάζονται για να αρρωγήσουν την Κομισιό σε διακυβερνητικό επίπεδο για τα θέματα υγείας και θεωρώ ότι έχουμε δώσει πολλά έγγραφα, έχουμε κάνει πολλές εργασίες για τη συμπερίληψη, την περιεκτικότητα, την αντιμετώπιση της ένδειας, των υπηρεσιών, τα θέματα της απασχόλησης. Αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε εργαστεί ποτέ για τα θέματα της υγείας. Δεν μας έχει απασχολήσει. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να δοθεί μια συνέχεια με πιο εύρωστο τρόπο για όλα αυτά τα θέματα από ό,τι μέχρι τώρα σε σχέση με το ερώτημα του αντίκτυπου της κρίσης για τα υγειονομικά συστήματα. Αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς. Μπορεί να έχουν γίνει κάποια πράγματα σε διμερές επίπεδο, αλλά παραμένει το θέμα της συλλογής δεδομένων στην Ευρωστάτ. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες και θα πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση, η δεύτερη παρατήρηση. Αναφερθήκατε στο θέμα της, ε, του εμβολιασμού. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε όλοι αν σκεφτόμαστε για μία έννοια ενός βασικού καλαθιού υγειονομικών υπηρεσιών που δεν θα πρέπει ποτέ να φύγουν, όπως είναι ο εμβολιασμό για ορισμένε ε, ασθένειε. Όπως μιλάμε για ελάχιστα κοινωνικά δικαιώματα, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να σκεφτούμε και για ελάχιστα υγειονομικά δικαιώματα. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πέσουμε κάτω από ορισμένα κατόφλια που περιλαμβάνουν ε, τη, τους εμβολιασμούς και άλλες βασικές υγειονομικές υπηρεσίες. Ένα τρίτο στοιχείο, το θέμα των ε, πληθυσμών που έχονται έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Γαλλία οι ξένοι πολλές φορές αντιμετωπίζονται με ικανοποιητικό τρόπο ακόμα, αλλά για τα άτομα που δεν έχουν ε, έγγραφα είναι τα πράγματα πολλές φορές πολύ αντικά. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ορισμένους στόχους που θα πρέπει να υλοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την περίθαλψη για τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με κάποιο ε, ομοιόμορφο τρόπο. Είπατε επίση και το θέμα, αναφερθήκατε για το θέμα τη συνολική κάλυψη, τη οικουμενική κάλυψη. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα στα άτομα τα οποία δεν βρίσκονται μέσα στο υγειονομικό σύστημα ασφάλιση να μπορούν να επωφελούνται από κάποια κάλυψη. Νομίζω ότι και αυτό είναι τμήμα των ε, θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν μεταξύ μα. Υπάρχει διαδικασία ελέγχου και ε, αξιολόγηση μέσω των ομοτήμων και αυτό μπορεί να γίνει πιστεύω ότι εκεί έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τα πράγματα. Πολλά μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η κρίση δεν θα είναι καταστροφή για όλα τα ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού και αυτό το έχουμε πετύχει στη Γαλλία σε κάποιο βαθμό. Σας ευχαριστώ. Κύριος ε, Ζεβελό. Ε, Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω δύο-τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Καταρχήν, θέλω να πω ότι έχουμε προετοιμάσει ένα κείμενο με συγκεκριμένες προτάσεις. Αν τα λέτε μπορούμε να σας το διαθέσουμε. Κατά δεύτερον, πράγματι υπάρχει μια αντιμεταρρύθμιση, ένα είδος αντιμεταρρύθμισης που τρέχει, δηλαδή σε ορισμένες χώρες και σε ορισμένους φορείς υπάρχει τόντι αυτή η τάση ε, να επανερχόμεθα στο παλιό ιατρικό μοντέλο ε, και στην παλιά αντιμετώπιση όσον αφορά άτομα με αναπηρία και άλλες ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας. Βέβαια, εμείς ε, πιστεύαμε ότι είχαμε φτάσει σε ένα σημείο όπου θα μπορούσαμε να βασίζουμε τις ε, δράσεις μας ε, και τις πράξεις μας στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλλον δεν ισχύει πια αυτό. Η νέα σύμβαση έφερε και μια νέα προσέγγιση στην αναπηρία. Η αναπηρία δεν είναι πρόβλημα του ατόμου, αλλά είναι ένα θέμα που έχει σχέση ανάμεσα την δική του την αδυναμία και τους φραγμούς που ε, προκαλεί η κοινωνία. Χωρίς τα γελιά μου δεν μπορώ να διαβάσω τις διαφάνειες. Αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε αντί να πηγαίνουμε πίσω στο μοντέλο των ε, ε, ελλείψεων πάντα σε σχέση με την απειρία. Τώρα, ας δούμε ποιο είναι το κόστος ε, του να μην επενδύσει κανείς σε, σε υπηρεσίες υγείας. Αυτή η ερώτηση που τέτοια είναι πάρα πολύ σημαντική. Το κόστος ε, της μη επένδυσης αφορά περισσότερο την απασχόληση, αφορά ε, τα μακροχρόνια επιδόματα. Το θέμα είναι να μπορεί κανείς να συμβάλλει στην κοινωνία και θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Μπορεί να ερωτηθεί κανείς πώς είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο σε μια χώρα της Κεντρικής Ευρώπης. Κάποια υπηρεσία έκλεισε για να μην κοστίζει. Και τι διαπιστώθηκε. Αν είχε παραμείνει για κάθε ευρώ επένδυσης θα προέκυπταν 16 ευρώ όφελος. Διότι η άνθρωποι θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην κοινωνία. Όμως ε, περικόπηκε αυτή η υπηρεσία. Και γιατί περικόπτουμε τέτοιου είδου υπηρεσίε. Αυτό είναι σημαντικό το ερώτημα. Και συμφωνώ μαζί σα ότι πράγματι υπάρχουν ε, δυνάμεις ε, στην κοινωνία που είναι αντιδραστικές και ίσως να υπηρετούν άλλους στόχους από το να αντιμετωπίζουν μόνο την κρίση. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Το είπα ήδη, ε, έχουμε εξετάσει το δυναμικό του τομέα για δημιουργία θέσεων απασχόλησης και αυτομάτως ο τομέας γίνεται τμήμα της λύσης και όχι του προβλήματος. Να βοηθήσουμε λοιπόν ε, τον κλάδο να επιτύχει κάτι και αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου, το Κοινοβούλιο μπορεί να εξετάσει και το νομικό πλαίσιο των νέων διαρθρωτικών ταμείων, τα οποία οφείλουν να προάγουν υπηρεσίες ε, που δίνουν δυνατότητες στους ανθρώπους και όχι να καταφεύγουν ε, όλοι στην ιδρυματοποίηση και στον διαχωρισμό των ανθρώπων της κοινωνίας. Το πακέτο κοινωνικών επενδύσεων πρέπει να είναι η σωστή προσέγγιση. Νομίζω λοιπόν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτή πρέπει να είναι η βάση των πράξεών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Γκούτουιν. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω και πάλι το τελευταίο σημείο. Νομίζω ότι όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την φροντίδα ατόμων με σοβαρές αναπηρίες περικόπτονται τώρα και αυτό αρχίζει να θίγει και θίγει βαθιά τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και έχουμε όλο το θέμα του ρατσισμού και των ανθρώπων που είναι μετανάστες οι οποίοι εργάζονται σε, στο χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο στην κοινωνία μας. Μία πάρα πολύ σημαντική συμβολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο διάλογο για το σεβασμό των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των διαφόρων ανθρώπων. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ ήμουν ένα ιδρυτικό μέλος μιας οργάνωσης φροντίδας στην Ιρλανδία και το μεγαλύτερο μέρος χρηματοδότησής μας έρχεται από επίσημες υπηρεσίες. Εμείς δεν βλέπουμε ο, να <coughs> μειώσουμε το ρόλο μας για να παροτρύνουμε τους δημόσιους φορείς. Και ο φορέας μας έχει ήδη υποστεί μια περικοπή 5 με 10% σε δημόσιους, ε, δημόσιους πόρους κάθε χρόνο τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως νομίζω ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις θα πρέπει να παρέχουν επιχειρήματα και να συνηγορήσουν υπέρ της προστασίας του ρόλου των φορέων που παρέχουν περιθέλψη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ Λίκη Πρόεδρος. Όλους τους και ευχαριστώ τους διερμηνείς οι οποίοι έμειναν μαζί μας μέχρι το τέλος. Ξέρω ότι η συγγήτρια θα καταθέσει και κάποιες προτάσεις στις 20 Φεβρουαρίου και θα την εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. is when it regards the pure health aspect. Here we will have to find out how we can, but it's internal business, but